Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά να λάβετε θέσεις για να αρχίσουμε αμέσως. Όπως θα ξέρετε, το, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε διερμηνία σε πάνω από 20 γλώσσες. Βλέπετε πόσες καμπίνες έχουμε στην αίθουσα. Είναι γεμάτες διερμηνείς και μπορείτε να παρακολουθήσετε διερμηνία στη μητρική της γλώσσα. Είναι πολύ βολικό αυτό και μας βοηθάει. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί μπορούμε όλοι να μιλάμε τη μητρική μας γλώσσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να καλωσορίσω δύο ε, εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, την κυρία Εύα που είναι πρόεδρος της Πολωνικής Βουλής, του ΣΕΙΜ και τον κύριο Μπορουσέβης που είναι πρόεδρος της Πολωνικής Γερουσίας. Θα συντονίσουν τις, τη συνεδρίαση αυτή ως συμπρόεδροι με συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε και εκπροσώπους από τα Εθνικά Κοινοβούλια, τους οποίους καλωσορίζω θερμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε τακτικά άπαξ το εξάμεινο τέτοιες ε, διακοινοβουλευτικέ ε, συνεδριάσει, προκειμένου να εξετάζουμε θέματα σημαντικά όπω τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα, πολύ σημαντική για όλου μα, φυσικά και την οικονομική κρίση που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο και τις κλιματικές αλλαγές. Ήταν τα θέματα των προηγούμενων τεσσάρων συνεδριάσεων, ε, κοινών συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά λοιπόν και τους ευρωβουλευτές μαζί με τους εθνικούς βουλευτές. Χαίρομαι ειλικρινά που βλέπω να καθόμαστε όλοι μαζί εδώ στην αίθουσα, Εθνικά Κοινοβούλια και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ε, καλωσορίζω και τον κύριο Μάικλ Τσίχον, που είναι ε, Διευθυντής Ασφάλειας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Εργασίας, στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας και αύριο θα έχουμε τον κύριο Βαντίσαφ Κοσίνιακ, που είναι πρόεδρος ε, εργασίας ε, και ε, κοινωνικής πολιτικής της Πολωνικής Βουλής, εκ μέρους του Συμβουλίου, και ο κύριος Λάσλο Άντορ, που είναι επίτροπος αρμόδιος για απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη. Θα λάβουν μέρος στην αυριανή πρωινή συνεδρίαση της κοινή κοινοβουλευτικής διάσκεψης. Α μην ξεχνάμε την υποχρέωση που μα δημιουργεί η συνθήκη τη Λισαβόνα να έχουμε όσο πιο τακτικέ επαφέ γίνεται. Είναι πολύ καλή αυτή η πρόταση και χαιρόμαστε για αυτή τη δυνατότητα που μα δίνει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Η συγκεκριμένη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση αφιερώνεται σε πολύ σημαντικά θέματα. Έχουμε τρία πάνελ, γνωρίζετε του τίτλου του. δεν χρειάζεται να σα του υπενθυμίσουμε. Ξέρετε ποια είναι τα αντικείμενα συζήτηση των τριών πάνελ. Μια όμως και ε, προτιμώ να μιλάω τη μητρική μου γλώσσα. Σας παρακαλώ να ακούτε αγγλικά, αλλά βάλετε τα ακουστικά σας, γιατί με βολεύει καλύτερα να μιλάω πολωνικά. Και θα περάσω στα πολωνικά και εγώ. Και πάλι λοιπόν, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Γερουσίας, αγαπητοί συνάδελφοι. Δύο χρόνια έχουν περάσει από τη θέση ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνας και είναι η πρώτη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλά για την αναγκαιότητα τακτικών επαφών, διακοινοβουλευτικών επαφών, δηλαδή επαφών μεταξύ των Εθνικών Βουλών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της δημοκρατικής μας ευθύνης τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγονται με παρόμοιο τρόπο, με άμεσες δηλαδή εκλογές, απευθείας από τους πολίτες. Και ευτυχώς που η συνθήκη της Λισαβόνας επισημαίνει την ανάγκη τέτοιων κοινών συνεδριάσεων. Έχουμε φυσικά ε, συνεδριάσεις και μεταξύ κοινοβουλευτικών επιτροπών, ε, στα πλαίσια της ΚΟΖΑΚ, όπως ξέρετε, στα πλαίσια των τη Ενάντησης Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να διαμορφώσουμε μία μεθοδολογία σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Αυτή η σκέψη είναι επίσης πολύ σημαντική και θα θέλαμε ε, να ενισχύσουμε αυτές τις πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ξέρετε, το σημερινό θέμα που πρότεινε η Πολωνική Προεδρία σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αντικείμενο της σημερινή συζήτηση ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό για τους συμπολίτε μας. Γιατί βρισκόμαστε σε κρίση, 116 εκατομμύρια απειλούνται με φτώχεια και ήδη 43 εκατομμύρια υποφέρει από πείνα, δηλαδή 8% του, του πληθυσμού της υπήρους μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να καταπολεμήσει τη φτώχεια και το λοιμό παντού στον κόσμο και είναι αδύνατο να διαφορήσει για ένα τέτοιο πρόβλημα ε, στο εσωτερικό της. Και φυσικά το ένα πολύ σημαντικό θέμα στα πλαίσια αυτά είναι η ανεργία, ιδιαίτερα των νέων, που σε ορισμένε περιοχέ ε, του Νότου ειδικά υπερβαίνει και το 40%. Μπορούμε να χάσουμε ολόκληρη γενιά δηλαδή με την ανεργία να μαστίζει τους νέους μας. Είναι σημαντικό λοιπόν οι ευρωπαϊκές πολιτικές και τα πολιετή δημοσιονομικά πλαίσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τα προγράμματα αυτά και τα πολιετή σχέδια μπορούμε να ε, μειώσουμε αυτή, αυτή την ανεργία 1,5 εκατομμύριο θέσει εργασία είχαμε χάρη στην πολιτική συνοχή μεταξύ του 2000 και του 2006. Ε, χάρη μόνο και μόνο στην πολιτική συνοχή δημιουργήθηκαν τόσε πολλέ θέσει απασχόληση και φυσικά έχουμε και τη γεωργική πολιτική. Ένα άλλο μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η γύραση του πληθυσμού. Τα επόμενα 30 χρόνια μέχρι το 2050 θα έχουμε διπλάσιο αριθμό ενηλίκων άνω των 60 ετών από τη σήμερα. Υπάρχει και το θέμα των ε, υπηρεσιών υγείας Φυσικά η μακροβιότητα είναι πολύ σημαντικό και πολύ θετικό θέμα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και υπογεννητικότητα και άρα αντιμετωπίζουμε δημογραφικό πρόβλημα. Γι' αυτό θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που προκαλούνται από τα συνδοξιδοτικά συστήματα. Γιατί και το θέμα της πρόορη δεξιδότησης θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν υπάρχει άλλη εναλλεκτική λύση. Θα πρέπει να δουλεύουμε περισσότερο, θα πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερες οικονομίες για να αποφύγουμε την υπερχρέωση. Δυστυχώ πολλέ χώρες σήμερα βρίσκονται υπερχρεωμένες και αυτά τα χρέη θα κληθούν να τα αποπληρώσουν οι επερχόμενες γενιές και αυτό είναι αντιδιοντολογικό. Δεν είναι ηθικό, δεν αρμόζει να επιρρύπτουμε το χρέος ε, στα παιδιά μας, ε, στα εγγόνια μας, στις επερχόμενες γενιές. Αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε από τώρα. Θα πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση. Θα πρέπει, όπως σας είπα, να παρατείνουμε το χρόνο ε, εργασίας, το συντάξιμο, την ηλικία εξόδου στη σύνταξη και αυτό ισχύει και για τις γυναίκες. Γιατί η ισότητα των ευκαιριών και η ισότητα των φίλων και η ε, υπόψη της ανάγκης πρόθεση μητρότητας, ώστε όλες οι γυναίκες που θέλουν να έχουν παιδιά να έχουν διευκολύνσει, γιατί όλες οι γυναίκες τελικά ανάλυση θέλουν να κάνουν παιδιά, να έχουν διευκολύνσει ώστε να μπορέσουν να συνδυάσουν τον οικογενειακό βίο, την προσωπική του ζωή με την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα ε, υιοθετήσαμε και ένα ψήφισμα για τις δημογραφικές γενιές και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τη γενετικότητα, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε ε, κατάλληλες συνθήκες εργασίας ε, και για τους ε, ενηλίκους άνω των 60 ετών. Να μην τους εξωθούμε δηλαδή στη σύνταξη και στην πρόορη σύνταξη μερικές φορές. Αλλά να τους επιτρέπουμε να εργάζονται περισσότερο. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα μας απασχολήσουν στην διάσκεψη αυτή. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες. Εγώ θα είμαι συνέχεια παρόν και το βράδυ θα έχουμε επίσημο δείπνο. Αύριο το πρωί θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις και θα ήθελα να υπογραμμίσω για μία, υπογραμμίσω για μία ακόμη φορά ότι η περίοδος της κρίσης μπορεί να είναι και ευκαιρία για να εγκρίνουμε κάποιες πολιτικές και κάποιες ε, ρηξικέλευθες ε, λύσεις και μεταρρυθμίσεις για πολλές πολιτικές όπως την οικονομική, την κοινωνική που χωρίς την κρίση δεν θα είχαμε την ευκαιρία. Αλλά αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Μερικές φορές σε ακραίες συνθήκες όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε άνευ προηγουμένου προκλήσεις πολύ συχνά καταφέρουμε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις και μάλιστα με πολύ σωστό και κατάλληλο τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουμε όλες αυτές τις πιθανές αλλαγές να δούμε μήπως χρειαζόμαστε νέα προσέγγιση για τις συντάξεις, για την αγορά εργασίας, για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, για την ενίσχυση της δημογραφικής ανάπτυξης. Για όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να συζητήσουμε, να εγκύψουμε σε όλα αυτά με καινοτόμο τρόπο. Και ίσως ε, η κρίση θα είναι ευκαιρία για κάτι τέτοιο. Αυτές ήταν σύντομες εισαγωγικέ παρατηρήσεις και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην ε, κυρία Εύα Κόπατς, στην πρόεδρο της Πολωνικής Βουλής, του ΣΕΙΜ, να της δώσω το λόγο γιατί θα ε, συντονίσει το επόμενο τμήμα της συζήτησης. Θα ήθελα καταρχήν, ε, κυρία Εύα Κόπετς, κυρία Πρόεδρε, να ζητήσω και από εσά κάποια εισαγωγικά σχόλια στη συζήτηση. Panie Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Πολωνικής Γερουσίας, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, κύριε και κύριοι Βουλευτέ, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Χαίρομαι ιδιαίτερω για την ευκαιρία που έχουμε για κοινή διακοινοβουλευτική συνεδρίαση ε, με συνδιοργάνωση της Πολωνικής Βουλής, της Πολωνικής Γερουσίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια της ε, κοινοβουλευτικής διάστασης ε, της Πολωνικής προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα είναι πραγματική τιμή Για μένα είναι πραγματική τιμή η έναρξη της 11 ε, ε, διακοινοβουλευτικής διάσκεψης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η παρουσία σα και η δέσμευσή σα δείχνει ότι η κοινοβουλευτική διάσταση έχει όλο και μεγαλύτερη διάσταση στην Ενωμένη Ευρώπη. Δυστυχώς αντιμετωπίζουμε μια κρίση και η διακοινοβουλευτική συνεργασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνδιοργάνωση τη σημερινή και αυριανή διάσκεψη. Η συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο τη κοινοβουλευτική διάσταση ε, τη Προεδρία Ευρωπαϊκή Ένωση Κυρίε και κύριοι, την 1η Δεκεμβρίου πέρασαν δύο χρόνια από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, ε, που δημιούργησε μια νέα θεσμική πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χάρη στην οποία τα εθνικά κοινοβούλια πολύ πιο ενεργά ε, παρακολουθούν την παρασκευαστική διαδικασία, συμμετέχουν ε, πιο δραστήρια σε αυτή. Ως θέλουμε να τηρηθούν οι αρχές της επικουρικότητας, ασκούμε ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο στο χώρο ασφάλειας, ε, δικαιοσύνης ε, και ελευθερίας, συμμετέχουμε στις αλλαγές μεταρρύθμισης της συνθήκης και πολύ πιο σημαντικό από όλα λαμβάνουμε ενεργό μέρος στην διακοινοβουλευτική συνεργασία. Τονίζω τη σημασία της τελευταίας αυτής συνεργασίας, γιατί ιδιαίτερα η συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλίων φέρνει πιο κοντά τους πολίτες, γιατί σε κοινοβουλευτικό φόρουμ έχουμε συζητήσεις για τα πιο σημαντικά θέματα που άπτονται του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδιαφέρουν άμεσα τους συμπολίτε μας. Η, σημαντική, η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή της ιστορίας της, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε την οικονομική κρίση που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ενωμένη Ευρώπη και αυτή η οικονομική κρίση απαιτεί από εμά όχι μόνο ε, υπεύθυνε αποφάσεις και αλληλέγγυα δράση, ταυτόχρονα όμως ε, μας υποχρεώνει να υιοθετήσουμε λύσεις που θα εξασφαλίσουν σταθερό και ήρεμο μέλλον στους πολίτες ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από τη στιγμή που θέλουμε η Ευρώπη να υλοποιήσει συγκεκριμένους ε, στόχους και να επανέλθει στο δρόμο της αηφόρου ανάπτυξης, θα πρέπει να εξετάσει διάφορες αλλαγές που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή κοινωνία και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις προκλήσεις των πολιτών στην Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. Γι' αυτό προτείναμε η σημερινή μας συνάντηση να αφιερωθεί σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Στην κοινωνική συνοχή και στην δημογραφική ανάπτυξη με υφόρο και ισορροπημένο τρόπο η διαδικασία της γύρασης του ευρωπαϊκού πληθυσμού συνεχίζεται. Γι' αυτό και η υπερβολική επιβάρηση των συνταξιδοτικών συστημάτων αποτελεί σημαντική απειλή για την ευημερία και την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη, ε, η οποία θέλουμε να χαρακτηρίζεται από συνοχή και ολοκλήρωση. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τις ε, για τα πολιτισμικά μας επιτεύγματα και ιδιαίτερα για τη μακροβιότητα των συμπολιτών μας. Γιατί αυτό οφείλεται στην βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, των κοινωνικών συνθηκών αλλά και των συνθηκών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην προσπάθεια υιοθέτηση πολύπλοκη πολιτική αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατεί να λειτουργήσει χωρί ε, ε, κοινωνία που θα χαρακτηρίζεται από συνοχή και ένταξη. Κάτι τέτοιο προποθέτει υψηλό επίπεδο απασχόληση, επενδύσει στι ειδικότητε και τι δεξιότητε, καταπολέμηση τη φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού και μάλιστα σε όλε τι περιφέρειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ιδιαίτερα σήμερα, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, σε τόσο χαλεπού καιρού για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να συνενώσουμε τι προσπάθειέ μα προκειμένου να περιορίσουμε τι ανισότητε σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη διαφόρων περιοχών και περιφερειών. Γιατί μια έλλειψη συνοχής ε, θα πρέπει να καταπολεμηθεί. Η κοινωνική συνοχή είναι σημαντική προτεραιότητα όχι μόνο της στρατηγική του 2020, αλλά και σημαντική έκφαση της αλληλεγγύης ε, στην Ενωμένη Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, στα πλαίσια της σημερινής μας ε, συνεδρίασης θα ήθελα να επικεντρωθούμε σε τρεις πολύ σημαντικές πτυχές και άξονες. Ο πρώτος είναι τα οικονομικά και δημοσιονομικά ζητήματα υπό το πρίσμα και των δημογραφικών αλλαγών. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι το θέμα της συνοχής στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης που θα είναι το αντικείμενο του δεύτερου πάνελ της διάσκεψης αυτής. Το τρίτο και τελευταίο πάνελ θα αφιερωθεί σε ε, κοινωνικά ζητήματα, ε, απασχόληση και δημογραφικές αλλαγές. Στη διάρκεια της συζήτησης ε, θα μπορέσουμε να δούμε ποιες είναι οι, που, ε, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε ό,τι αφορά τη δημογραφική ανάπτυξη στη σύγχρονη Ευρώπη. Γιατί απέναντι σε μια οικονομική κρίση το πρόβλημα αυτό της δημογραφικής ε, ανάπτυξης οξύνθηκε και λύση θα πρέπει να αναζητούμε ήδη από σήμερα. Έχω πάντως την ελπίδα και την αίσθηση ότι και η σημερινή συνάντηση και τα συμπεράσματά της ε, δεν ε, θα σταματήσουν εδώ, αλλά θα δοθεί συνέχεια και θα συμβάλλουν στην δημογραφική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί από τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης θα εξαρτηθεί όχι μόνο το μέλλον των δικών μας, αλλά και το μέλλον των επερχόμενων γενναιών. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία και ας μεριμνήσουμε για το κοινό ευρωπαϊκό μας πεπρωμένο. Πιστεύω ότι η σημερινή μας συνάντηση, ε, μάλιστα σε τόσο χαλεπούς ε, καιρούς και σε τόσο δεινή οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση, θα συμβάλλει ε, στην συζήτηση για την κοινωνική συνοχή και τη δημογραφική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε της Πολωνικής Βουλής. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που σίγουρα καλύπτουν όλο το φάσμα της σημερινής συζήτησης και χαίρομαι που οριοθετήσατε τόσο σαφώς τους τρεις άξονες της συζήτησης και τα τρία πάνελ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην επόμενη μιλήτρια. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Κόπετς για να δώσει το λόγο στον κύριο Μάικλ Τσίχων, που είναι διευθυντή ε, του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Σα ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σα και σας δίνω το λόγο, κύριε Μάικλ Τσίχων. Thank you, Madam President. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, μέλη της Πολωνικής Βουλής και Γερουσίας και μέλη των άλλων Εθνικών Κοινοβουλίων εξ ονόματο Διεθνού Γραφείου Εργασία. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπούζεκ και την κυρία Κόπατ για την ευκαιρία να προσφωνήσω του ε, ευρωβουλευτέ και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου από τα κοινοβούλια των κρατών μελών στην αίθουσα και να παρουσιάσω τι απόψει του Διεθνού Γραφείου Εργασία για τι δημογραφικέ αλλαγέ και τι επιπτώσει στην κοινωνική συνοχή <clears throat> ακριβώς όσον αφορά την ενεργοποίηση της ε, Ευρώπη Αλληλεγγύης. Ζητήθηκε να δώσω μια σύντομη εισαγωγή στα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα και αύριο. Και αυτό που θα κάνω θα είναι τρία πράγματα. Πρώτον, θα ανακεφαλαιώσω κάποια σημαντικά στοιχεία για τις δημογραφικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους. Μετά θα αναφερθώ στις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές και στις εντάσεις και στο τέλος θα παρουσιάσω τις πολιτικές επιλογές που ταυτοποιούνται από μια πρόσφατη δημοσίευση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για τις Δημογραφικές Αλλαγές. Θα προσπαθήσω να τα κάνω όλα αυτά και μια και έχω μόνο 10 λεπτά ταχύτατα θα τα καλύψω. Πρώτον, Όσον αφορά κάποια στοιχεία, κάποια είναι γνωστά, κάποια άλλα είναι λιγότερο γνωστά. Και ίσως ε, αυτό είναι κάπως, ε, μας εκπλήσει κάπως. Όλοι γνωρίζουμε τις ε, περιβόητες καμπύλες που αυξάνονται κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημίσεως του προηγούμενου αιώνα μέχρι το 2010 στην Ευρώπη λιγότερο σημαντικό από τη συστημική συνολική το ποσοστό εξάρτησης, δηλαδή του αριθμού των παιδιών και εκείνων που πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες τους από τους ε, εργαζόμενους ε, που ε, έχουμε ένα ποσοστό 60% και αυτό είναι το σχετικό μέγεθος των μετατροπών και μεταμορφώσεων που πρέπει να επιτύχει η κοινωνία στην Ευρώπη για να καλυφθούν οι ανάγκες των εξαρτημένων μελών. Φαίνεται υψηλό αυτό το ποσοστό, αλλά δεν είναι τόσο υψηλό όσο τα δημογραφικά ποσοστά. Και έχουμε και τις πιέσεις όσον αφορά το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδοτήσεων. Και αυτό ακριβώς ε, παρουσιάζει η Ευρώπη σήμερα. ποσοστά που βλέπουμε ότι ε, υπάρχει υπεργύρανση και υπάρχει μείωση των ε, εργαζομένων. Θα υπάρξει αυτή η ένταση μέχρι το 2010 και σε κάποιες χώρες πολύ περισσότερο. Ταυτόχρονα η ε, ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξηθεί και σαν αποτέλεσμα, και αυτό μας εκπλήσει, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σύνολο των δημοσίων δαπανών στο σύνολο της Ευρώπης θα αυξηθεί λόγω της υπεργύρασης κατά 4,6% του ΑΕΠ μεταξύ σήμερα και του 2016. Δηλαδή κατά ένα περίπου μία ποσοστία μονάδα ανά δεκαετία. Κάποιες χώρες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις τεράστιες αλλαγές. Το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Ωστόσο, δεν ε, βαίνουν εκ παραλίλου οι οικονομικές εξελίξεις. Έχουμε τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και της ε, κρίσης και είναι πιθανόν ότι θα οδηγηθεί η κατάσταση στο να μειωθεί η απασχόληση, να συρρυκνωθεί η απασχόληση τις επόμενες δεκαετίες. Δεκαετίες μεταξύ 2020-2050 κατά το ίμιση. Τα ποσοστά που είδαμε στο παρελθόν μέχρι το 2010 δεν θα ε, μπορέσουν να επιτευχθούν. Πρέπει να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και πρέπει να την δούμε έναντι της ε, συνολικής μείωσης κατά 1,5% του ΑΕΠ από το 1998 μετά από δεκαετίες διαρκούς αύξησης βλέπουμε ότι ο ανταγωνισμός, φορολογικός ανταγωνισμός μπορεί να είναι ένα από τα αίτια. Ταυτόχρονα όμως όσον αφορά το ποσοστό του ΑΕΠ μειώνεται συνολικά στην Ευρώπη έχουμε απώλεια από 1,5-1,6% από τις αρχές του 2000 και από το 1970 που υπήρχε σχετική αύξηση βλέπουμε αυτή την ε, μετάθεση μετατίθεται το θέμα από τους μισθούς ε, όσον αφορά την ε, κερδοφορία και το συνολικό κόστος ε, της εργασίας μέσω του ανταγωνισμού και μέσω της παγκοσμιοποίησης μπορεί να είναι ένα πιθανό αίτιο αυτής της κατάστασης. Τι έχουμε ως αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων και πιέσεων. Αν επεκτείνουμε τις σημερινές πολιτικές και τη σημερινή ανακατανομή πλούτου ε, στο μέλλον, ε, αν τίποτα δεν αλλάξει, θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλο και μεγαλύτερη πίεση ανταγωνισμού με συρρυκνούμενο πληθυσμό, ενεργό πληθυσμό. Και έτσι θα είναι λιγότερο παραγωγική αν τίποτα δεν αλλάξει. Θα λιμνάσουν τα ποσοστά ανάπτυξης ε, ή θα οπισθοχωρήσουν και θα συνεχίσει να μειώνεται το ΑΕΠ λόγω του ανταγωνισμού και θα υπάρξει ε, αποτελμάτωση όσον αφορά και τα φορολογικά έσοδα. Βλέπουμε ότι το ποσοστό ε, σε σχέση με τον ε, ενεργό πληθυσμό και του άνεργου πληθυσμού θα είναι πραγματικά δυσμενές. Ο ανταγωνισμός αυτός έχει αυτές τις επιπτώσεις. Συνολικά το επίπεδο διαβίωσης ή θα επιδεινωθεί ή θα οπισθοχωρήσει ή θα αποτελματωθεί. Και βλέπουμε ότι αυτό έχει αρνητικότατες επιπτώσεις στους εργαζόμενους αυξανόμενα βάρη για τους ε, εξαρτώμενους και την οικογένεια θα οδηγήσει σε μια υποχρεωτική ανακατανομή σε σχέση με τις γενναίες και μέσα, στην ίδια, την, ε, ε, μέσα σε μια ίδια γενναία βλέπουμε ότι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά μπορούν να θεωρηθούν δείκτες ε, για μια κατάσταση που αν δεν αλλάξει θα χάσει τη μάχη η Ευρώπη. Τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει αυτή η εξέλιξη και πρέπει να δούμε ότι έχει μειωθεί και το ποσοστό ανάκτησης των απολειών και όλα αυτά είναι περαιτέρω ενδείξεις ότι η αλληλεγγύη συρρυκνώνεται και αυτή η κοινωνική αλληλεγγύη. Το σύστημα κοινωνικής προστασίας, η εχμή του δόρατος κατά το παρελθόν της κοινωνίας στην Ευρώπη που είχε δημιουργήσει την κοινωνική συνοχή γίνεται τώρα πεδίο μάχης με τις προσαρμογές στις νέες εξελίξεις. Δείχνουν όλα αυτά μια επιδίνωση του κοινωνικού ιστού. Η πρόοδος αυτή είναι σταδιακή, όμως ε, βρίσκεται υπό εξέλιξη και δυστυχώς πολλοί συνταξιούχοι ε, ζουν τα πάνδυνα, βιώνουν τα πάνδυνα εδώ και αρκετό καιρό. Και βλέπουμε για τις εναλλακτικέ πολιτικές ε, πολλοί από εμά δεν, θα δεν θα αντιμετωπίσουν ήρεμα κάποιες από αυτές. Έχουμε κάποιες επιλογές και θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε όλες. Ο βαθμός εξάρτησης όσον αφορά την κοινωνία θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα βιώσιμο επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό. Γενναίες χωρίς παιδιά ή με λίγα παιδιά πρέπει να μπορούν να παραμείνουν ενεργές επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να είναι παραγωγικές μέχρι ότου οδηγηθούν στην ε, συνταξιοδότηση. Αυτό όμως δεν είναι πανάκια δεν θα μπορέσει διαφορετικά η κοινωνία να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της μόνο αυξάνοντας το επίπεδο ε, συνταξιοδότησης, την ηλικία συνταξιοδότησης. Πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν. Τα καθεστώτα χρόνου εργασίας πρέπει να θεσπιστούν παράλληλα με αξιοπρεπείς όρους ε, απασχόλησης. Δίκαιες πολιτικές μετανάστευσης πρέπει να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν. Και πάλι όμως αυτά δεν είναι πανάκια. και οι υιοθετούν ή μιμούνται τις ε, αναπαραγωγικές τάσεις ε, και προσανατολισμούς της ε, κοινωνίας υποδοχής. Όλα αυτά μπορούν να είναι συμβατά με αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν ή υποθέτουμε ότι θα είναι η εξέλιξη της κοινωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παραγωγικότητα θα πρέπει να βελτιωθεί, να υπάρξουν μεγάλε επενδύσει στην εκπαίδευση και την παιδεία για να μπορέσει να προετοιμαστεί το ανθρώπινο δυναμικό να είναι παραγωγικό. Επενδύσεις στην διαβίω εκπαίδευση πρέπει να γίνουν και να διασφαλιστούν θέσει απασχόληση για του ε, ε, υπερήλικου που θα πρέπει και εκείνοι να μπορούν να βρουν μια θέση εργασία και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ε, ε, εργασιακής τους ζωής όταν ε, η υγεία τους έχει υποστεί επιδείνωση πλησιάζοντας την, το όριο συνταξιοδότησης. Πρέπει και οι όροι διαβίωσης και οι όροι εργασίας να είναι συμβατοί με αυτές τις εξελίξεις σε σχέση με την αγορά εργασίας. Και τέλος, δεν είναι το τέλος, αλλά εν πάση περιπτώσει πολιτικές θα πρέπει να δημιουργηθούν που θα αντιμετωπίζουν όπως αναφέρθηκε και στην δυνατότητα ανάκτησης του ποσοστού γεννητικότητας ώστε να μπορέσουν οι οικογένειες να ανταποκριθούν, να ανταπεξέλθουν μέσα σε ένα πλαίσιο πιο φιλικό για αυτές όπου η περίθαλψη και η φροντίδα καθώς και η εκπαίδευση και η παιδεία θα την χάνουν υψηλής προτεραιότητας θα πρέπει να δούμε τις επιπτώσεις ε, που έχουν ε, όλοι αυτά, όλα αυτά τα στοιχεία στην ε, ζωή των εργαζομένων μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας. Υπάρχουν κλασικές συνταγές που είναι πολύ καλά γνωστές σε σχέση με την χρήση της οποίας την χάνουν. Όλα αυτά όμως στις περισσότερες φορές θα πρέπει να δούμε ότι θα συνεπάγονται δαπάνες, ιδιαίτερο κόστος, το οποίο πρέπει τώρα να καλυφθεί και δεν θα είναι καθόλου ε, χαμηλό αυτό το επίπεδο κόστους ε, οι δαπανών. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθηθούν αυτά τα μέτρα από πολιτικές, ε, οικονομικές και φορολογικές. Πρέπει να υπάρξει μια νέα σχέση ΑΕΠ σε σχέση με την φορολογία και να μην υπονομευθούν οι στόχοι μας. Κάποιες ε, από τις ε, οικονομίες της Ευρώπης ε, έχουν ένα τέτοιο υψηλό ποσοστό χωρίς απώλεια ανταγωνισμού. Μόνο αυτά τα μέτρα θα δημιουργήσουν ένα δίκαιο πλαίσιο ανακατανομής πλούτου που χρειάζεται στην Ευρώπη για να υπάρξει ένα δίκαιο καθεστώς και ένα πάγιο ισχυρό καθεστώς επενδύσεων που θα οδηγήσει σε πρόοδο. Οδηγούμε στα συμπεράσματα. Η υπεργύρανση, η γύρανση είναι για τα άτομα μια ευλογία. Είναι όμως δαπανηρή αυτή η διαδικασία και αποτελεί πρόκληση για τις κοινωνίες μας και είναι και μια παγκόσμια αναγκαιότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί για να αντιμετωπιστούν ε, προβλήματα και στενοποί και να υπάρξει μια δίκαιη αντιμετώπιση των ε, ηλικιωμένων. Πρέπει να ε, δούμε αυτή την εξέλιξη προς την γύρανση και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και της ανακατανομής πλούτου. Η αλλαγή συμπεριφοράς και η αλλαγή ακριβώς της σύνθεσης των κοινωνιών μας είναι ένα πρόβλημα. Οι Ευρωπαίοι θέλουν και ε, πρέπει να συνεχίσουν να ζουν σε ένα καθεστώς ε, ειρηνικής συμβίωσης. Και παρόλα τα προβλήματα θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να γίνουν πιο παραγωγικοί χωρίς ε, να υπονομευθεί ο κοινωνικός ιστός. Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην παιδεία και την εκπαίδευση στους ε, μαθητές στην εκπαίδευσή τους, να υπάρξει ένας τρόπος εξέβρεσης δίκαιας κατανομής του πλούτου όσον αφορά τα εισοδήματα των πολιτών. Θα πρέπει να πληρώνονται και υψηλότερα ποσοστά φόρων. Θα πρέπει να δεχθούμε και το γεγονός της μετανάστευσης και έτσι να αντιμετωπίσουμε την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Αυτό που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις και αυτές τις αλλαγές. Και εν τέλει θα μπορούσα να συμπεράνω ότι μακροπρόθεσμα, ότι οι πολιτικές αυτές που χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμα μπορούν να εφαρμοστούν στην Ευρώπη υπέρ των πολιτών σε σχέση με τα εισοδήματα, τους μισθούς και την κοινωνική προστασία. Και όλα αυτά από κοινού μπορούν να επιτευχθούν αν οι σύνθεση του κοινωνικού ιστού και των πολιτικών της Ένωσης σταματήσει, μπορέσει να αναχαιτιστεί και μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό του μισθολογικού κόστους μέσα σε μια κοινωνία που γυράσκει όλο και περισσότερο. Να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε τις απώλειες με κοινωνική συνοχή. Ευχαριστώ. Dziękuję panu Cichoniowi za wystąpienie. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας δώσω κάποιες πληροφορίες. Μαζί με τον πρόεδρο της Γερουσίας, τον κύριο Μποροσέβιτς, ε, θα συντονίσουμε και το, δεύτερο, θα συντονίσει το δεύτερο πάνελ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Σρέντερ και στον κύριο Έτμουντ Βίτπροντ, ε, που θα είναι η συμπρόεδρη του πρώτου πάνελ. Ja, einen schönen Μάλιστα, καλό σας απόγευμα σε όλους σας. Για μένα είναι η πρώτη ε, φορά, η πρώτη αυτή ευκαιρία να συμμετάσχω με αυτόν τον τρόπο και να βρίσκομαι εδώ πάνω ανάμεσά σας και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την ευκαιρία. Θέλουμε τώρα να περάσουμε στο πρώτο πάνελ οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα και επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής των δημογραφικών αλλαγών. Πολλοί έρχονται από περιφέρειες και περιοχές ε, που πλήττονται ιδιαίτερα και γνωρίζουν από τα βιώματά τους το τι συμβαίνει. Λόγω της ευημερία ε, γυράσκει όλο και περισσότερο πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει αναφερθεί και το γνωρίζουμε. Συρρυκνώνεται όμως επίσης ο πληθυσμός και σε κάποιες περιοχές υπάρχει μία μελέτη για τις ε, περιοχές και περιφέρειες ε, του 2020 υπάρχει ένα κεφάλαιο για αυτό το θέμα. Σε κάποιες περιφέρειες όλο και πιο έντονο θα είναι το φαινόμενο αυτό, διότι υπάρχει αποψήλωση του πληθυσμού, οι νεότεροι φεύγουν από αυτές τις περιφέρειες και επαρχίες, πάνε όλο και περισσότερο στα αστικά κέντρα λόγω αστιφιλίας. Ποιες ε, προσεγγίσεις υπάρχουν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τέτοιων περιοχών που αποψηλώνονται λόγω αστιφιλίας. Εγώ προέρχομαι από μια περιοχή που βρίσκεται πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα και είναι το, η περιοχή, η επαρχία με τα μεγαλύτερα, με το μακρύτερο σύνορο προς την Πολωνία. Και μετά υπάρχουν δύο φιλοσοφίες. Η μία φιλοσοφία λέει να αφήσουμε στη φύση αυτές τις περιφέρειες και με προγράμματα για τον τουρισμό να δείξουμε πόσο όμορφη είναι η φύση σε αυτές τις περιφέρειες και περιοχές και να ανακερδιθεί, να ανακτηθεί η φύση. Η δεύτερη φιλοσοφία, φιλοσοφική προσέγγιση λέει να μην εγκαταλείψουμε αυτές τις περιφέρειες και επαρχίες, να διατηρηθούν οι υποδομές, ε, να διαφυλαχθούν και να προετοιμαστούν για να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες προκλήσεις της αστιφιλίας και αποψήλωσης. Προσβλέπουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας. Ο κύριος Τσαβίνσκι πρώτος θα δώσει μια εισαγωγή. Πού βρίσκεται? Εσείς κύριε Τσαβίνσκι εκεί. Μάλιστα, είσαστε ο εισηγητής εσείς και έχετε προετοιμάσει ένα κείμενο ως εισαγωγή. Παρακαλώ να μας το παρουσιάσετε σύντομα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσαβίνσκι και το λέω αυτό σύντομα, από το 2005 είναι στην ΣΕΙΜ, στην Πολωνική Βουλή. Προέρχεται από την πόλη Νόβα Σάς και από το 1994 μέχρι το 2000 ήταν δήμαρχος εκεί από την χριστιανοδημοκρατική πλατφόρμα ε, κομματικού σχηματισμού που εκφωνήθηκε στα πολωνικά και ο διερμηνέας δεν μπόρεσε να κρατήσει. έχει τον λόγο παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, εγκαινιάζοντας τη συζήτηση αυτή με θέματα τόσο σημαντικά ζητήματα και προκλήσεις που μας παρουσίασε προηγουμένως και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Γεζιμπούς και ε, Μπουζέκ, η Πρόεδρος της Πολωνικής Βουλής, η κυρία Κόπατς, αλλά και ο Πρόεδρος του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ο κ. Τσίχων, θα ήθελα να θέσω μερικά ερωτήματα, κάποια ερωτήματα που στη διάρκεια της ε, σημερινής συζήτησης θα αναλυθούν, θα ρίξουν λίγο φως στο μέλλον και θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα να υποβάλουμε στο πάνελ μας κάποιες συστάσεις για το τι μέλη γενέστε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Καταρχήν, υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα ή όχι. Σε αυτή την ερώτηση ήδη έχουμε απάντηση. Το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ρητά και κατηγορηματικά ότι το δημογραφικό πρόβλημα είναι υπαρκτό και θα πρέπει να το επιλύσουμε. Με ποιο τρόπο όμως. Γιατί αν αφήσουμε το πρόβλημα να αυτορυθμιστεί μόνο του, να αφήσουμε αυτό το ζήτημα στο, στο έλεος του, με κίνδυνο να ε, ή να ε, περιοριστεί, τι θα γίνει, ή θα διωγκωθεί, ή, θα, δεν θα διωγκωθεί, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα, ή θα διωγκωθεί όμως, οπότε θα αντιμετωπίσουμε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Νομίζω ότι στόχος μας είναι να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση προκειμένου να υλοποιήσουμε το στόχο μας. Και ποιος είναι ο στόχος αυτός. Στόχος της δικής μας δραστηριότητας θα πρέπει να είναι η αναζήτηση της σταθερότητας, ε, της σταθερότητας για τις επερχόμενες γενιές. Και αν προγραμματίσουμε <coughs> κάποιες εργασίες και κάποιες δραστηριότητες που οι στατιστικολόγοι και οι εμπειρογνώμονες ήδη έχουν προετοιμάσει, γιατί η διάγνωση έχει γίνει, γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα. Το δημογραφικό πρόβλημα, η γύραση του πληθυσμού, η υπογεννητικότητα, το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης, τα δημοσιονομικά προβλήματα, να αυξηθεί η φορολογία, να μειωθούν οι συντάξεις ε, να αναλυφθούν κάποιες αναπτυξιακές προσπάθειες προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν διευκρινιστεί, έχουν απαριθμιστεί και έχουν ιεραρχηθεί ανάλογα με τη σημασία τους. Οπότε ανακύπτει το ερώτημα. Όλα αυτά τα ζητήματα ε, πώς θα τα ε, αντιμετωπίσουμε και πώς θα θέσουμε σε εφαρμογή τις λύσεις. Ποιος θα πρέπει να βρει τις λύσεις και να τις εφαρμόσει. Κάθε χώρα χωριστά, κάθε χώρα ξεχωριστά υπολογίζοντας στα δικά της ατού και στα δικά της πλονεκτήματα ή μήπως τα προβλήματα αυτά θα πρέπει να επιληθούν σε κεντρικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια λύση θα είναι η πιο βιώσιμη και η πιο σταθερή. Πολλές φορές ε, αναφέρεται ότι όταν ε, το βάρος επιμερίζεται σε πολλούς χάνει τη βαρύτητα του και γίνεται πιο ελαφρύ. Αυτό ίσως αυτή είναι και η λύση ε, στην Ευρώπη να δούμε επιτόπου πού υπάρχει το πρόβλημα σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε περιοχή και σε κάθε χώρα και να προσπαθήσουμε όλοι από κοινού για να εξασφαλίσουμε ένα σταθερό μέλλον στην Ευρώπη και να αναλάβουμε και την προσωπική του ευθύνη ο καθένας. Γιατί αυτά τα ζητήματα τα έχουμε εντοπίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά να γνωρίζουμε ταυτόχρονα και την ιδιαιτερότητα τη κάθε περιφέρειας και την πολυμορφία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε περιοχή έχει δικά τη ατού ιδιαιτερότητε και προτερήματα. Αν αυτά τα προτερήματα τα συνδυάσουμε και κάθε περιοχή ε, αξιοποιώντας τα προσπαθήσει να βρει λύσεις, και ο καθένας αναλάβει το μικρό του φορτίο σε δικό του επίπεδο, τότε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αποτέλεσμα θα είναι πιο ορατό. Οπότε ανακύπτει και το άλλο ερώτημα. Έχουμε το χρόνο για κάτι, νομίζω, για κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι η απάντηση εδώ είναι σαφής. Έχουμε ακόμη ε, λίγα χρόνια για την προετοιμασία των λύσεων και για την εφαρμογή τους. Αν όμως δεν ξεκινήσουμε από τώρα ήδη να ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά, θα πανικοβληθούμε γιατί θα μείνουμε πίσω και τελευταία στιγμή θα προσπαθήσουμε σπασμωδικά να βρούμε λύσεις. Η δημογραφική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή, η ισορροπημένη Ευρώπη, η φόρος ανάπτυξη, όλα αυτά τα προβλήματα που μας απασχολούν σήμερα είναι σημαντικές προκλήσεις. Ε, για αυτές μπορούμε να δείξουμε σε μια διετία ότι περάσαμε τις εξετάσεις και πραγματικά αξιοποίησαμε την ευκαιρία για συνεργασία και κοινή δράση. Ευχαριστώ. Ähm, Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Τσαβίσκη για αυτή τη σύντομη εισαγωγή σε αυτό το θέμα. Και τώρα θα ήθελα να, να πω σύντομα ότι για, εμείς για τους διάφορους εθνικούς βουλευτές και τους ευρωβουλευτές έχουμε μια κάποια σειρά που θέλουμε να τηρήσουμε. Δύο εθνικοί βουλευτές ε, και ε, ένας ευρωβουλευτής, ένα λάξ, να έχουμε μια, ένα καλό μείγμα παρεμβάσεων από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις παρεμβάσεις και κάθε βουλευτής θα έχει μόνο τρία λεπτά στη διάθεσή του για την παρέμβασή του για μια σύντομη τοποθέτηση δήλωση και με το ρολόι θα παρατηρούμε, θα υποπτεύουμε ερωτώ τώρα ποιοι θέλουν να παρέμβουν έχουμε και κατάλογο, έχουμε πίνακα εδώ ωραία, έχουμε κατάλογο για τις παρεμβάσεις έχουν προαναφερθεί οι, όσοι θα παρέμβουν και τώρα από τους σοσιαλδημοκράτες ο κύριος Κέρλοφ θα λάβει τον λόγο. Ο κύριος Κυρίλοφ. Δεν παρήσατε όμως ο κύριος Κυρίλοφ. Και θα έλεγα να πάρουμε τους επόμενους που θέλουν να παρέμουν. Εθνικός βουλευτής από την Assemblée Nationale, από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ο κύριος Ζακ Λενάη, παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ στις συνέπειες της οικονομικής και της δημοσιονομικής της δημογραφικής αλλαγής. Η Γαλλία όπως και άλλες χώρες γυράσκει σύμφωνα με τις προβλέψεις του 2010 της στατιστικής υπηρεσίας και αν δεν αλλάξει κάτι η Μητροπολιτική Γαλλία θα έχει 73.600.000 κατοίκους το 2060, δηλαδή 11 εκατομμύρια περισσότερους από ότι το 2007. Ο αριθμός αυτών που είναι άνω των 60 θα αυξηθεί κατά 10 εκατομμύρια, δηλαδή το 2060 ένα στους τρεις Γάλλους θα είναι άνω των 60. Τρεις παράγοντες παίζουν ρόλο. Η αύξηση του προσδόκιμου, το λεγόμενο baby boom, και ένα επίπεδο γεννητικότητας χαμηλότερο από το ποσοστό αντικατάστασης των γενεών. Αυτό επηρεάζει φυσικά τους δημοσίους λογαριασμούς και τα κοινωνικά ταμεία. Σε μακροοικονομικό επίπεδο η γύρανση αυτή έχει επιπτώσεις δύσκολα μετρήσιμες στο δυναμικό ανάπτυξης. Πέραν του επίπεδου δυνητικής ανάπτυξης, τα αποτελέσματα της γύρανσης της δημογραφικής θα επηρεάσουν την συνέχεια του γαλλικού συστήματος κοινωνικής κάλυψης. Η γύρανση προκαλεί προβλήματα στις ε, μεταφορές ανάμεσα στις γενναίες. Οι μεταφορές αυτές είναι προς δύο κατευθύνσεις, από τους νέους προς τους ε, ε, γυράσκοντες προς τα πάνω, μέσω δημοσίων ταμείων, μέσω χρηματοδότησης ε, των συντάξεων και επίσης και προς τα κάτω μέσω των κληρονομικών δικαιωμάτων. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν αυτές το 18%. Ενώ στο μέλλον αυτό το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί. Το οικονομικό βάρος θα επιβαρύνει τους νέους. Βλέπουμε ότι δεν θα υπάρχουν πλέον υψηλού επίπεδου προς τα κάτω μεταφορές πιστώσεων και αυτό κινδυνεύει να οδηγήσει σε ένα πόλεμο γενεών. Μία αντικαταστατική σε εισαγωγικά μετανάστευση θα ήταν άραγε σε θέση να διατηρήσει τη δημοκρατική ισορροπία και τον ενεργό πληθυσμό. Τίθεται το θέμα αλλά υπάρχουν αμφιβολίες. Τα μεταναστευτικά ρεύματα μέσω ειδικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων αυξάνουν αυτούς που πληρώνουν εισφορές, αλλά τελικά δεν επηρεάζουν το σύνολο των συντάξεων και τον αριθμό των αδρανών πολιτών. Η Γαλλία το 1993, το 2003 και μετά το 2008 αλλάζει συνεχώς την πλήρη συνταξιοδότηση. Αυτές οι τρεις μεταρρυθμίσεις εφαρμόστηκαν δύσκολα, αλλά παρόλα αυτά μείωσαν το έλλειμμα το οποίο περιμένουμε για το 2050. Αλλά από ό,τι φαίνεται η Γαλλία τα επόμενα χρόνια πρέπει να κάνει περαιτέρω προσπάθειες για να περιορίσει το κόστος και το ποσοστό των συντάξεων στα πλαίσια του ΑΕΠ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε. Στη συνέχεια Ο κύριος Κέβιν Χόπκινς από τη Μεγάλη Βρετανία, από το House of Commons, την Βουλή των Κοινοτήτων. Εδώ παρίσταται. Yeah. Μάλιστα. Ωραία. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Thank you, Madam Chair. Um, and, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να πάρω το λόγο Μιλάμε για τον γυράσκοντα πληθυσμό και τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται. Έχουμε ανάγκη και από πολύ περισσότερους νεοτέρους για να συντηρήσουν τους μεγαλύτερους στην Ιταλία. Παρ' όλα αυτά εμείς στην Μεγάλη Βρετανία έχουμε προβλήματα γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που δεν έχουν δουλειά, εργαζόμενοι επίσης που συνταξιοδοτούνται και θέλουν να δουλέψουν περισσότερο δεν μπορούν να το κάνουν. Υπάρχει ένα πρόβλημα λοιπόν. Έχουμε πολύ περισσότερους πρόθυμους να εργαστούν και δεν έχουμε τις θέσεις εργασίας που είναι απαραίτητες. Αν είχαμε πλήρη απασχόληση θα είχαμε πολύ υψηλότερους φόρους, θα είχαμε μειότερο θα έλεγα έλλειμμα και θα αντιμετωπίζαμε την κατάσταση που αντιμετωπίσαμε στην εποχή του baby boom με ανάπτυξη και ευημερία για όλους. Πρέπει λοιπόν το πρόβλημα της μαζικής ανεργίας να αντιμετωπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν μπορώ να πω τώρα πώς θα πρέπει να γίνει αυτό βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ένα επιμέρους θέμα, το θέμα της της ιδιοκτησίας στις προχωρημένες ηλικίε ξέρουμε ότι οι συντάξεις μειούνται, οι ιδιωτικές εταιρείες δεν παρέχουν συστήματα συνταξιοδοτικής κάλυψης, τα παρεχόμενα από την ελεύθερη αγορά δεν είναι ε, αποτελεσματικά και πάρα πολλοί εργαζόμενοι δεν βλέπουν πώς θα καλύψουν τις ανάγκες τους σε προχωρημένη ηλικία. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα σύστημα υποχρεωτικό κρατικό που να συνδέεται με τις αμοιβέ των εργαζομένων για τη συνταξιοδότησή τους αν θέλουμε να καλύψουμε τις ανάγκες του γυράσκοντα πληθυσμού και να πείσουμε και τις επιχειρήσεις ότι κάτι τέτοιο είναι θετικό. Δύο επιμέρους σημεία. Συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σισόν και η ανάλυση του. Κάποια από τα συμπεράσματά του ίσως δεν με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο, αλλά η ανάλυση του είναι πάρα πολύ σωστή. Μιλήσατε και για την ανάγκη αύξησης του ποσοστού των γεννήσεων. Δεν ισχύει αυτό για μας το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε υψηλότατο επίπεδο γεννήσεων και έχουμε αυξάνοντα αριθμό πληθυσμού. Το θέμα είναι ε, έχει ενδιαφέρον. Έχουμε πάρα πολλούς, σαν παράδειγμα και στην εκλογική μου περιφέρεια, Πολωνούς, οι οποίοι οι πολωνικής καταγωγής που γεννούνται εκεί και κτλ. Δεν είναι αυτή η λύση λοιπόν. Βέβαια ζητώ συγγνώμη γιατί εγώ έδειξα τα προβλήματα, δεν έδειξα τις λύσεις, θα χρειαζόμουν δύο ώρες για να το κάνω. Ίσως οι συνάδελφοι μπορούν να σας βοηθήσουν. Ένα συνάδελφος τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τους σοσιαλδημοκράτες. Ο κύριος... Σκυλακάκης. Όχι, συγγνώμη, ο κύριος Σκυλακάκης από τους φιλελεύθερους. Ο κύριος Θεοδωρός Σκυλακάκης, παρακαλώ. Είναι στην αίθουσα, ελπίζω. Μάλιστα. Ωραία. Έχετε τον λόγο κύριε Σκυλακά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, οι δημογραφικές εξελίξεις είναι πράγματι μια πολύ μια πολύ δύσκολη πρόκληση γιατί δεν συμβαίνουν μόνο εντός Ευρώπης αλλά και εκτός Ευρώπης. Έχουμε ένα πληθυσμό που γυράσκει στην Ευρώπη και έναν πολύ μεγάλο πληθυσμό που θα αυξηθεί πολύ περισσότερο εκτός Ευρώπης και θα διεκδικήσει και πόρους και αγορές ε, σε παγκόσμιο επίπεδο περιμένουμε μέχρι το 2050 περίπου 2 δισεκατομμύρια ακόμη ανθρώπους τουλάχιστον να μπουν στην παγκόσμια αγορά. Είναι λοιπόν διπλή η πρόκληση. Στο εσωτερικό της Ευρώπης δεν υπάρχουν πολύ εύκολοι τρόποι για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Είμαστε υποχρεωμένοι είτε να δουλέψουμε παραπάνω είτε αυτοί που δουλεύουν να παράγουν πολύ περισσότερο για να μπορούν να ζήσουν στο ίδιο επίπεδο οι περισσότεροι ηλικιωμένοι που θα έχουμε μπροστά μας. Συνεπώς πρέπει να κινηθούμε σε πολλά επίπεδα. Ασφαλώς πρέπει να διευκολύνουμε την εργασία και σε μεγαλύτερη ηλικία. Σε πολλά κράτη-μέλη είναι πολύ δυσκολότερο να εργαστείς όσο περνούν τα χρόνια και κοινωνικά αλλά και από πλευράς κινήτρων και συνταξιδοτικών συστημάτων αυτό είναι λάθος. Ε, οι άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι είναι σε όλο και καλύτερη φυσική και πνευματική κατάσταση σήμερα και πάρα πολλοί επιθυμούν να συνεχίσουν να δουλεύουν. Το δεύτερο είναι στα ίδια μας τα ασφαλιστικά συστήματα να κοιτάξουμε πολύ περισσότερο την έννοια των ορισμένων εισφορών αντί για τις ορισμένες παροχές. Να μπορούμε δηλαδή να οργανώνουμε τα ασφαλιστικά συστήματα με βάση τις εισφορές που καταβάλουν οι ασφαλισμένοι και όχι με βάση ε, αυτά που θα επιθυμούσαν το πολιτικό σύστημα να τους δώσει γιατί αυτό πια δεν είναι διατηρήσιμο και οι προσαρμογές που πρέπει να γίνουν υπερβαίνουν την πολιτική ικανότητα των περισσότερων ευρωπαϊκών πολιτικών συστημάτων και το βλέπουμε αυτό και στις χώρες του Νότου καθώς είναι υποχρεωμένες υποχρεωμένα τα πολιτικά συστήματα σήμερα να μειώνουν τις συντάξεις, ε, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο πολιτικά. Και το τρίτο επίπεδο παρεμβάσεων αφορά την υγεία. Η υγεία είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί όσο περισσότερο ηλικιωμένοι είναι οι άνθρωποι τόσο αυξάνεται το κόστος του υγειονομικού συστήματος. Και εκεί πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος στην πρόληψη και στον τρόπο ζωής. Είναι ανάγκη να επενδύσουμε σε αυτά τα επίπεδα και να το κάνουμε αυτό και πανευρωπαϊκά. Δεν έχουμε αντιληφθεί όσο θα έπρεπε τις οικονομικές συνέπειες του τρόπου που λειτουργούν τα συστήματα υγείας που στηρίζονται κυρίως ε, στα φάρμακα και στην μετά την ασθένεια επέμβαση ως σήμερα. Ε, τελειώνω λέγοντας ότι υπάρχει πολλή δουλειά και οι λύσεις είναι και ευρωπαϊκές, όχι μόνο εθνικές. Ευχαριστώ. Πολύ χαιρόμαστε που το ακούμε αυτό από ένα Ευρωβουλευτή. Τώρα έχουμε και τους ε, αγορητές που θα προετοιμάζονται ε, είχα πει λόγω του ότι η οθόνη ανέφερε κάποιον που είχε ήδη παρέμβει και έτσι δεν αλήθευε αυτή η σειρά. Τώρα από την Γερμανία ο κύριος Ράινχαρτ ε, Πίζεκ έχει τον λόγο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τον λόγο. Είμαι όμως από το Αυστριακό Κοινοβούλιο και όχι από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, ζητώ συγγνώμη. Ε, εξαρτώμαι από τα σημειώματα που μου δίνουν οι βοηθοί και είχε ε, εσφαλμένα αναφερθεί ότι είσαστε από τη Γερμανία, ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη, σφάλμα ήταν και δεν είναι καθόλου ε, υποεκτίμηση του ε, ατόμου σας, καθόλου δεν σας ε, περιφρονούμε. Από την Λέντα ε, Κάμερ είσαστε, από το σώμα των ε, κρατηδίων από την Αυστρία ο κύριος Ράινχαρτ Πίσετς λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα της δημογραφικής αλλαγής που δεν μπορεί όμως να εξεταστεί μεμονωμένα όσον αφορά και τις οικονομικές εξελίξεις και για την χρηματοδότηση των δημογραφικών αλλαγών. Αν πάρουμε ένα παράδειγμα από την Αυστρία, στην Αυστρία υπάρχει ακραία με, ε, διαφορά σε σχέση με την πραγματική ηλικία που προβλέπεται από τον νόμο για την συνταξιοδότηση 59 έχουμε ως ε, έτος ε, συνταξιοδότησης και πρέπει να αλλάξει αυτό το πλαίσιο γιατί από πλευράς χρηματοδότησης έχουμε φτάσει στα όρια της αντοχής μας και πρέπει να δούμε και την ε, επανένταξη των ε, ηλικιωμένων στην ε, αγορά εργασίας. Και έχουμε και το θέμα της μείωσης και των μισθολογικών βαρών και των παρακολουθημάτων όσον αφορά την μισθολογική επιβάρυνση όσον αφορά και τις ε, εισπράξεις, ε, ε, τις εισφορές των εργοδοτών. Θα πρέπει να μπορούν οι εργοδότες να μπορούν να απασχολούν και ηλικιωμένους εργαζομένους. Και με τη σειρά πρέπει να τα πάρουμε και να δούμε ότι πρέπει να κινήσουμε από την χρηματοδότηση που στην Αυστρία πάνω από ένα τέταρτο του συνολικού προϋπολογισμού χρηματοδοτείται από τους φόρους μισθών, μισθολογικής, ε, μισθωτής εργασίας. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι διαφέρω από την προηγούμενη παρέμβαση που έγινε ότι εδώ καλείται το κράτος να δράσει. Το κράτος πρέπει να δημιουργήσει το δημόσιο της προϋποθέσεις ώστε οι εργαζόμενοι και οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι να μπορούν να επανέρχονται στην αγορά εργασίας και να επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας. Το κράτος πρέπει να ανακουφίσει, να δημιουργήσει προγράμματα ελάφρυνσης ε, όσον αφορά την επανένταξη και εργασία των ε, ηλικιωμένων. Δεν είναι δυνατόν τα μισθολογικά βάρη και η φορολογία να είναι υπερβολικά ε, όσον αφορά τους ε, ηλικιωμένους εργαζόμενους. Ε, όσον αφορά την μισθωτή εργασία και την φορολογία, στην Αυστρία έχουμε δύο, εκατομμύρια που βλέπουμε ότι επιβαρύνονται ιδιαίτερα και πρέπει σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό να ληφθεί υπόψη λόγω της οικονομικής κρίσης και των ε, Τη βεβαρημένη κατάστασης. Καλείται το κράτος λοιπόν να δράσει, να δημιουργήσει τι προϋποθέσεις και όρου ώστε οι εργαζόμενοι να βρουν την οδό προς την κοινωνική επανένταξη και εργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέγει η πρόεδρο, τώρα έχουμε έναν εκπρόσωπο από το Κοινοβούλιο της Κύπρου, από την Βουλή της Κύπρου. Ο κύριος Χρήστος Τηλιανίδη, λοιπόν παρακαλώ έχει τον λόγο. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Yes. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας φέρνω την εμπειρία από μια μικρή χώρα η οποία είναι ανάλογη και μάλλον ακριβώς ίδια με τις εμπειρίες ολόκληρης της Ευρώπης και επειδή αναγνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα ότι είναι κοινό αναμφισβήτητα πρέπει να ξεκινήσουμε από κοινέ λύσεις. Γι' αυτό θα συμφωνήσω με τη θέση ότι χρειάζονται ευρωπαϊκές πολιτικές, κατά κύριο λόγο και μετά οι εθνικές πολιτικές που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, είναι το πρώτο, που σημαίνει ότι μέσα στη γενικότερη κρίση της Ευρωζώνης και γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποία, με την, στην οποία ψάχνουμε να βρούμε καινούργια εργαλεία οικονομικής πολιτικής ευρωπαϊκής θα πρέπει να εντάξουμε και τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης και τα θέματα του δημογραφικού προβλήματος. Το ένα είναι αυτό, ότι χρειαζόμαστε κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές. Το δεύτερο είναι ότι, και υπόθηκε και αυτό και θέλω να το ενισχύσω, είναι ότι χρειάζεται να αυξήσουμε τα όρια συνταξιοδότησης, τα όρια ηλικία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Από τη στιγμή που αυξήθηκε το προσδόκιμο ζωής, πρέπει αναπόφευκτα να πάμε και σε αύξηση των ορίων ηλικία συνταξιοδότηση. Α μην φοβηθούμε το πολιτικό κόστο. Εδώ πρέπει να εντάξουμε και τη φιλοσοφία του flexibility, τη ευέλικτη εργασία που θα πρέπει να συμπεριλάβει και τα άτομα τρίτη ηλικία που θα μείνουν στην αγορά εργασία. Και το τρίτο που θέλει μια περισσότερη ριζοσπαστικοποίηση των θέσεων και απόψεών μας είναι όντως η ενσωμάτωση μέρους του μεταναστευτικού ρεύματος. Δεν πρέπει να το φοβηθούμε. Έχουμε δυνατότητες να κάνουμε αυτή την ενσωμάτωση με ένα αποτελεσματικό και υγιή τρόπο και πρέπει να το επιχειρήσουμε. Νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει κοινή αποδοχή του προβλήματος, κοινή αναγνώριση, πρέπει ως πολιτικά όντα να μπούμε στις προτάσεις. Και οι προτάσεις να είναι συγκεκριμένες στη βάση αναλογιστικών μελετών γιατί η αριθμοί όπως έχει δείξει και την τελευταία κρίση στην οικονομία και σε αυτά τα θέματα είναι αμήλικτοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μία συνάδελφος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η κυρία Ντανούτα Γιασλοβιέσκα. Ντανούτα Γιασλοβιέσκα, παρακαλώ. Ζοβιέτσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι αναφιβολό ότι όταν συζητούμε για τα δημογραφικά προβλήματα θα πρέπει να έχουμε υπόψη την δραστηριοποίηση στην αγορά εργασίας. Σήμερα η κινητικότητα που είναι από τις πρωταρχικέ και θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, είναι σε πολύ χαμηλό ποσοστό. Μόνο 2% των Ευρωπαίων πολιτών εργάζονται σε χώρα διαφορετική από την πατρίδα τους και 17% δηλώνει ότι θα ενδιαφερόταν να εργαστεί σε άλλο, σε άλλο κρατός μέλος και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχουμε πολλά παραδείγματα και τα συζητάμε με τους συναδέλφους. Ε, στην ε, Βαβαρία υπάρχει έλλειμμα 500.000 εργαζομένων. Ε, Επίση έχουμε την Πολωνία, τη Τσεχία, τη Σλοβακία, στη Γαλλία έχουμε αύξηση της ανεργίας. Είναι δύσκολο να αξιοποιηθεί αυτό το εργατικό δυναμικό που πολύ συχνά είναι υψηλά εξειδικευμένο, έχει διεξιότητες, αλλά δεν μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα κινητικότητας. Μερικές φορές επίσης υπάρχει ε, μικρή πρόσβαση σε πληροφορίες για την διαθεσιμότητα αυτών των θέσεων απασχόλησης. Άλλος λόγος είναι η εξαιρετικά διαφοροποιημένη κοινωνική πολιτική στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν τόσες διαφορές ε, μεταξύ των κοινωνικών πολιτικών και ο κόσμος ε, δεν γνωρίζει τι να περιμένει, ποια είναι τα δικαιώματά του. Επίσης υπάρχει αδιαφάνεια στα συνταξιδοτικά συστήματα. Οι νέοι προσπαθούν με πολύ ε, όριμο τρόπο να σχεδιάσουν το μέλλον τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις ε, και το τέλος τη επαγγελματική του σταδιοδρομία και προσπαθώντα να προγραμματίσουν και τη σύνταξή του. Γι' αυτό και χρειάζονται τις πληροφορίες. Χρειαζόμαστε λοιπόν πολλές προσπάθειες και σε επίπεδο παιδεία, εκπαίδευση. Και εκεί διαπιστώνουμε ότι στην ε, Ευρώπη χρειαζόμαστε ρηξικέλευθες αλλαγέ και σε θέματα παιδεία. Έχουμε ελάχιστου ε, νέου με τεχνικέ δεξιότητε. με βασικές ειδικότητες και πολλές φορές χρειαζόμαστε τέτοιους τεχνικούς και ανειδικευτούς εργάτες. Επίσης, ελάχιστα προετοιμάζουμε τους νέους μας για μια ε, ελαστικότητα και για ένα άνοιγμα και για μια καλύτερη προσαρμογή στις συνθήκες εργασίας, ώστε να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα προβλήματα που θα εμφανιστούν στην πορεία της σταδιοδρομίας τους. Μιλούμε για την αγορά εργασίας. Υπάρχει ένα γεφύρωτο χάσμα μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και των ε, ε, ανθρώπων που αναζητούν μια θέση απασχόλησης. Γιατί ε, παρακολουθούμε την αγορά εργασίας σε υψηλό επίπεδο, αλλά δεν παρακολουθούμε άμεσα την κατάσταση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενώ σε τελική ανάλυση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που εξασφαλίζουν τις περισσότερες θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κοινωνικό ταμείο που αξιοποιούμε για να ε, ενισχύσουμε το εργατικό δυναμικό ε, και πάλι ελάχιστη είναι η συμβολή του. Ε, δυστυχώς ε, μερικές δεκάδες χιλιάδες είναι οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται και όχι εκατοντάδες χιλιάδες όπως τα περιμέναμε και θα χρειαζόμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μπορώ να τα πω αυτά γιατί κατάγομαι από μια χώρα που πολύ αποτελεσματικά αξιοποιεί τα κονδύλια του κοινωνικού ταμείου. Σίγουρα υπάρχουν τρόποι για να αξιοποιήσουμε καλύτερα το κοινωνικό ταμείο, κάτι που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών για να εξασφαλίσουμε καλύτερη αξιοποίηση. Και δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση. Νέε θέσει απασχόληση δημιουργούν όχι μόνο οι υφιστάμενε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και οι νέοι που μπορούν ανεξάρτητα να ασκήσουν ένα ελεύθερο επάγγελμα. Για τέτοιους νέους αυτοαπασχολούμενους υπάρχει έλλειψη κεφαλαίου, υπάρχει έλλειψη πρόσβαση στο κεφάλαιο, δεν υπάρχουν αρκετές, ε, ε, αρκετές, ε, αρκετά μέτρα για να μπορέσουν να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους και έτσι δεν μπορούν να ούτε να δημιουργήσουν θέσει απασχόληση για του ίδιου, ούτε να δημιουργήσουν θέσει εργασία και για άλλου. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να βρούμε λύσει. Να καλύψουμε αυτέ τι αδυναμίε που εντοπίζουμε στην αγορά εργασία. Γιατί υπάρχει δυνατότητα αυτέ τι αδυναμίε να τι διορθώσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Τώρα, στη συνέχεια, ένα αγορητή από τη Γερουσία τη Πολωνία, ο κύριο Μάρεκ Ζιογόφσκι. Παρακαλώ. Σα Σας ευχαριστώ για την ε, τιτάνια αυτή προσπάθεια να, προσφέρετε, να προφέρετε σωστά το όνομά μου. Σε ό,τι αφορά τι δημοσιονομικέ συνέπειε των δημογραφικών αλλαγών, θα ήθελα να πω ότι αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο ε, δίλημα. Ε, για πολλά χρόνια καταναλώναμε και ξοδεύαμε πολύ περισσότερα αυτά που παραγάγαμε και αυτό, αυτή, αυτό οδήγησε στην κρίση του κράτους πρόνοιας, γιατί το κράτος πρόνοιας ήταν από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ε, Ευρώπης και του ευρωπαϊκού μοντέλου, αλλά αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί, γιατί έχουμε αφενός ένα γεράσκοντα πληθυσμό, που αφενός αποτελεί ευλογία και επιτυχία, αλλά ο γεράσκοντα πληθυσμός απαιτεί περισσότερες δαπάνες και ε, μας έχει φέρει σε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε τις δαπάνες, ενώ ταυτόχρονα διανύουμε μια οικονομική κρίση που απαιτεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ε, πειθαρχία. Η, η δημογραφία είναι μια επιστήμη πολύ ακριβής και σαφής. Γνωρίζουμε τι θα συμβεί μετά από 50 χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε και τη λύση και μάλιστα με πνεύμα αλληλεγγύης. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να επιφέρουμε τις απαραίτητες αλλαγές έχοντας υπόψη και τις επερχόμενες γενές, γιατί ξέρουμε ε, τι θα συμβεί ε, μέσα σε 20 χρόνια. Δεν θέλουμε λοιπόν το βάρος των δράσεών μας και ιδιαίτερα τις αδράνειές μας να το επιρρύψουμε στους ώμους των παιδιών και των εγγονιών μας. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο λοιπόν. Όχι μόνο ανάγκη ε, δημοσιονομική πειθαρχία και λιτότητας, αλλά χρειαζόμαστε και οικονομική ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο της αλληλεγγύης αν επιφέρουμε κάποιες αλλαγές, το βάρος θα πρέπει να επιμεριστεί σε όλες τις ομάδες που μπορούν να αναλάβουν αυτό το, βάρος. Ομάδες, οργανώσεις, γιατί μερικές τράπεζες λέμε ότι παρά είναι ε, μεγάλες για να αποτύχουν. Ενώ άλλοι παράγοντες είναι πολύ φτωχοί για να έχουν την πολυτέλεια να πληρώσουν τις ε, μεταρρυθμίσεις αυτές. Αλληλεγγύη λοιπόν και αυτό και χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό όχι μόνο για τη δημοσιονομική πειθαρχία των ε, ε, ευρωπαϊκών χωρών, αλλά θα πρέπει να έχουμε καλύτερη, καλύτερο συντονισμό και των ευρωπαϊκών κοινωνικών πολιτικών. Νομίζω ότι ο κύριος Μπούζεκ στην αρχή της ε, συνεδρίασης είπε μια πολύ σωστή φράση. Είπε ότι ε, βρισκόμαστε σε κίνδυνο με την οικονομική κρίση, αλλά η κρίση θα μπορούσε να είναι και ευκαιρία και κίνητρο για να κινητοποιηθούμε. Να δώσουμε ενάψματα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να κάνουμε και κάποιες θυσίες στις μακρο, μακροπρόθεσμες πολιτικές και χάρη σε αυτή την κρίση να δράξουμε την ευκαιρία και να μπορέσουμε να κρατήσουμε και την αισιοδοξία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στον πίνακά μου, μια και στην οθόνη ίσως είναι διαφορετικά, έχω εδώ μια, μια βουλευτή γυναίκα. Είναι πολύ καλό ότι μια γυναίκα τώρα θα, θα παρέμβει. Από το Λετωνικό Κοινοβούλιο, η κυρία Σατακαλίνιδα. Λουκασιέβιτσα. Ελπίζω ότι βρίσκεται στην αίθουσα. Δεν το πρόφερα σωστά το όνομά σα. Έκανα λάθο. Η κυρία Λουκασέβιτσα, παρακαλώ. Εντάξει, τώρα έχουμε έναν άλλο κατάλογο. Δεν παρίσταται λοιπόν. Εντάξει. Και τώρα έχουμε κάποιον από το Τσεχικό, από την Βουλή της Τσεχίας, από το Κοινοβουλευτικό Σώμα, από την Βουλή. Η κυρία Τσαλαμκόβα, παρακαλώ. Γιτκα Τσαλαμκόβα. Η κυρία Γίτκα Τσαλαμκόβα, παρακαλώ. Καλό σα απόγευμα, καλή σα μέρα, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτά και βρίσκω ότι στον γύρο μιας κοινή συζήτησης θα έπρεπε να αναφερθεί αυτό ως άποψη. Ακούσαμε ότι χωρίς τη μετανάστευση θα αποθάνει η Ευρώπη, θα αποβιώσει η Ευρώπη. Κάνουμε λόγο εδώ για τα προβλήματα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, τα προβλήματα της ευημερίας, του κράτους ευημερίας, που καλύπτει τις περισσότερες ανάγκες και λειτουργίες μιας οικογένειας, την περίθαλψη και φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων κτλ. Τώρα θα πρέπει να αναγνωριστεί η αξία της εργασίας για να έχει και η γυναίκα τον μισθό της και να εισπράττονται και εισφορές. Θα πρέπει τα μέσα αυτά αμέσως μετά τη γέννηση ενός παιδιού να μπορούν να, οι γυναίκες να επιστρέφουν μετά τη γέννηση, την γένα στην αγορά εργασίας. Πολλές φορές ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, εντάσεις και τριβές όσον αφορά και την οικογενειακή ζωή και την επαγγελματική ζωή και αυτό οδηγεί πολλές φορές στο να μειώνεται το ποσοστό γεννητικότητας και βλέπουμε ότι δεν είναι πλέον δυνατό να διατηρηθεί με αυτόν τον τρόπο και να χρηματοδοτηθεί η κοινωνία του κράτους ευημερία. Και οι οικογένειες όλο και περισσότερα ε, καθήκοντα πρέπει να καλύπτουν και να επιτελούν το, θα, της εργασίας και την ανάληψη υποχρέωσης περίθαλψης και φροντίδας ηλικιωμένων ταυτόχρονα, καθώς και πολυσχηδεί πολλά, ε, πολλαπλά καθήκοντα. Το κράτος ε, οδηγεί στο να επομίζονται αυτά τα βάρη. Το κοινωνικό κράτος όμως και η επιστροφή στην αγορά εργασίας ε, χρειάζονται μία μετάθεση. Μετά από την γέννηση ενός παιδιού οι γυναίκες πρέπει να επιστρέφουν στην αγορά εργασίας. Βλέπουμε ότι δεν υποστηρίζονται τέτοια μέτρα όμως σε μεγάλο βαθμό υπάρχει μια κοινωνία που γυράσκει, ε, γίνεται όλο και πιο υπερήλικη και δεν υποστηρίζονται πλέον ε, οι οικογένειες παρότι είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας μας. Γι' αυτό θα πρέπει να τεθούν προτεραιότητες, να δοθούν προτεραιότητες, προτεραιότητα στην οικογένεια, να υποστηρίξουμε τις οικογένειες με τέτοιο τρόπο ώστε η οικογένεια να μπορεί να επομίζεται τα καθήκοντά της και να τα υλοποιεί με το σωστό τρόπο. Πρέπει υποστηρικτικά να μπορέσουμε να δράσουμε το κράτος πρέπει τις διαφορετικές δυνατότητες προσφοράς ε, να δράσει το κράτος για την περίθαλψη και φροντίδα των ηλικιωμένων. Είναι σημαντική η εκστρατεία ενημέρωσης και πληροφόρησης. Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε ότι η κοινωνική συνοχή έχει το επίκεντρό της, την έδρα της στις οικογένειες. Και από εκεί ξεκινά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τώρα στον συμπρόεδρο κύριο Edmund Wittbrod να δώσω τον λόγο στον κύριο Wittbrod για την ε, πρωτοκαθεδρία που θα αναλάβει των εργασιών στη συνεδρίασή μας. Ελπίζω θα τα καταφέρει καλύτερα από μένα και ως πρόεδρος της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Πολωνικής Γερουσίας. Είναι πολύ καλό το ότι βρισκόσαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα αναλάβετε τώρα τα ενία αυτής της συνεδρίασής μας. Παρακαλώ. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, γερουσιαστή Μιετσίσουαφ Ογκούστη από την Πολωνική Γερουσία. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο θέματα. Το πρώτο αφορά την πολιτική... Διακόπτε, συγγνώμη, το μικρόφωνο. Η πολιτική ε, θα πρέπει να έχει ε, πολυσύνθετο και οριζόντιο χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τομείς που αποτελούν ε, αρμοδιότητα και των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλες ε, οι πολιτικές θα πρέπει να καλύπτονται. Η, πολιτική, η αναπτυξιακή πολιτική, η καινοτομία... Ε, η πολιτική για θέματα υγείας και ούτω καθεξής. Επίσης, θα πρέπει η πολιτική να καλύπτει όλους τους φορείς, όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πολιτική, τις, α, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί αυτοί εφαρμόζουν εμπράκτως σε περιφερειακό επίπεδο την πολιτική αλλά και τους εθνικούς α, φορείς. Γιατί οι πολιτικές αυτές ε, είναι υποχρεωτικές ε, και για τα κοινωτικά θεσμικά όργανα και για τα εθνικά και για τα περιφερειακά όργανα. Γιατί αν κατακαιρματίσουμε την προσπάθεια δεν θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε στη σημαντική αυτή πρόκληση. Θα πρέπει με συνεργασία να την αντιμετωπίσουμε. Έρχομαι και στο δεύτερο θέμα τέθηκε μία ερώτηση. Μήπως μας απειλεί ο πόλεμος μεταξύ των γενεών. Καλό θα ήταν να εμβαθύνουμε σε αυτό το ζήτημα, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος για τέτοιος πόλεμος μεταξύ των γενεών. Γιατί θα... μπορεί να γίνει πόλεμος για τις θέσεις απασχόλησης και για τα χρήματα, γιατί χρειάζονται χρήματα για την επιβίωση, αλλά και για την ανάπτυξη των διαφόρων γενεών. Μερικές φορές ε, ε, ακούγεται μια θεωρία που δεν στηρίζεται από τις μελέτες και τις έρευνες ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτε σε πολωνικό επίπεδο γιατί έχουμε ε, πολωνούς ε, επιστήμονες που επιβεβαιώνουν ότι δεν ισχύει ότι οι ηλικιωμένοι που παραμένουν στην αγορά εργασίας κλέβουν τις θέσεις εργασίας από τους νέους. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό είναι ένας μύθος. Γιατί όσο ε, περισσότερη ε, απασχόληση υπάρχει στους ηλικιωμένους, τόσο μικρότερη ανεργία υπάρχει και στους ε, νέους. Φαίνεται ότι η παραμονή στη θέση εργασίας των ηλικιωμένων είναι ένα κίνητρο για πρόσβαση, καλύτερη πρόσβαση εργασίας και των νέων. Πώς γίνεται αυτό. Καταρχήν, μειώνεται η πίεση στο συνταξιοδοτικό σύστημα με την παράταση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Και έτσι μειώνεται το κόστος της εργασίας και αυξάνεται ταυτόχρονα η ανταγωνιστικότητα. Εφόσον υπάρχει μια εξορρόπηση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, βελτιώνεται ταυτόχρονα και η οικονομική και η δημοσιονομική κατάσταση των κρατών. Και έτσι ε, πολύ περισσότερα κονδύλια μπορούν να τα αφιερώσουν στην ανάπτυξη. Φέτος ε, η Πολωνία για όλα τα εξοδοτικά συστήματα θα χρειαστεί ε, να πληρώσει 94 δισεκατομμύρια ζώτη από τους φόρους. Αν, αυτά τα, αυτά, αυτές τις δαπάνες μπορούσε να τις, αυτά τα κονδύλια να τα αφιερώσει στην αναπτυξιακή πολιτική, Σίγουρα η οικονομική της ανάπτυξη ήταν πολύ μεγαλύτερη και άρα θα δημιουργούνταν πολύ, πολύ περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ της παραμονής των ηλικιωμένων στη, ε, στην αγορά εργασίας και άρα στην παράταση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και ε, στην ανέβρεση, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για τους νέους. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Ας μην φοβηθούμε λοιπόν και ας μην δηλιάσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γερουσιαστά Αουγκουστίν. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο James Κλάπισον από την Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο ότι το θέμα της απασχόλησης είναι το καθοριστικό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε όλη την Ευρώπη και επίσης να δούμε πώς θα μπορέσουμε να πληρώσουμε την ε, απόσυρση από την αγορά εργασίας ενός γυράσκοντα πληθυσμού. Ακούστηκαν από ορισμένου ομιλητέ ότι υπάρχει έλλειψη νέων ανθρώπων. Δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε έλλειψη θέσεων απασχόλησης για του νέους. Έχουμε ένα εκατομμύριο άεργους νέους και έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες νέους στο Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα κατάρτισης και οι προοπτικές για αυτούς είναι πραγματικά ιδιαίτερα σκοτεινές και φοβάμαι ότι θα έχουμε να κάνουμε στο μέλλον αν δεν αλλάξουν τα πράγματα με ένα γενεακό πρόβλημα που θα οδηγήσει σε περαιτέρω περιπλοκές. Έχουμε εκατομμύρια ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, οι οποίοι μαζί με τους αέργους έχουν μια πολύ θα έλεγα επιπόλαια σχέση με την αγορά εργασίας και είναι στα όρια του να είναι ανενεργοί ε, εργασιακά. Το θέμα δεν είναι ότι χρειάζονται κάποια μικρά μαθήματα ή κάποια περαιτέρω κατάρτιση αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει και μια προκατάληψη για ανθρώπους οι οποίοι περνούν μια κάποια ηλικία και υποτίθεται δεν έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν στην παραγωγή. Θα πρέπει όμως να αλλάξουμε την οτροπία και να βρούμε θέσεις εργασίας για αυτούς τους ανθρώπους. Εκεί που διαφωνώ με αυτά τα οποία άκουσα, όπως επίσης και με τον κύριο Κισό, να πω ότι στην περίπτωση του Ενωμένου Βασιλείου η μετανάστευση δεν είναι το αποτέλεσμα. Μπορεί να είναι καλό πράγμα, μπορεί να βοηθάει τις οικονομίες ανάλογα στη φάση στην οποία βρίσκονται. Αλλά νομίζω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο το θέμα της συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας και της κάλυψης των κοινωνικών ασφαλίσεων το θέμα δεν είναι η έλλειψη προσώπων αλλά και η υπερβολική παρουσία μερικές φορές προσώπων και η μετανάστευση αυτή είναι ένα πρόβλημα. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μετά τη Γερμανία τη μεγαλύτερη παρουσία μεταναστών και σε έδαφος μικρότερο από το αντίστοιχο γερμανικό. Και θα φτάσουμε σε λίγα χρόνια, ίσως και σε 70 εκατομμύρια κατοίκους, οι οποίοι θα μένουν κυρίως, θα είναι συμπυκνωμένος, θα έλεγα, ο πληθυσμός αυτό στην ανατολική πλευρά και στην Αγγλία. Σας ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε της Βουλής των Κοινοτήτων. Τώρα θα λάσω το λόγο στον κύριο Ίγμαρ Νίλσον από τη Σουηδική Βουλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, μιλήσουμε όχι μόνο για το δημογραφικό πρόβλημα, γιατί ε, μιλούμε για το δημογραφικό πρόβλημα σαν να ήταν ε, κάτι αρνητικό, σαν να ήταν ένα πρόβλημα. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε υπό ένα θετικό πρίσμα, να θεωρούμε τη δημογραφική ανάπτυξη ως μια θετική εξέλιξη. Βέβαια, τα συνταξιοδοτικά συστήματα στηρίζονται στην εμπιστοσύνη, στην εμπιστοσύνη μεταξύ των γυναιών. Αν πληγεί αυτή η εμπιστοσύνη, τότε θα δημιουργηθεί κρίση στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, πριν από 20 χρόνια εγκαινιάσαμε ένα νέο συνταξιοδοτικό σύστημα που δεν ανήκει, δεν εμπίπτει στον προϋπολογισμό γιατί κυρίως στηρίζεται σε προκαθορισμένες συνδρομές και όχι σε προκαθορισμένα ωφέλη. Και είναι πολύ πιο ελαστικό το σουηδικό σύστημα. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο, μπορεί κανείς ε, να εργαστεί όσο θέλει και τα χρόνια εφαρμογή αυτού του συστήματο, του νέου συστήματο, διαπιστώσαμε ότι ο μέσο όρο ηλικία ε, συνταξιοδότηση έχει αυξηθεί κατά δύο χρόνια. Δεν φανταζόμασταν ότι η εξέλιξη ήταν τόσο ραγδαίε. Ήταν πολύ θετικέ, παρόλο που είναι δύσκολο να τι διαχειριστεί κανεί. Ακόμη και στη Σουηδία αντιμετωπίζουμε προβλήματα και τα προβλήματα οφείλονται κυρίως στην έλλειψη χρηματοδότησης γιατί όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν αυτό το σύστημα. Όσο μειώνεται η απασχόληση, τόσο μειώνονται τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση του συνταξιδοτικού συστήματος. Πολύ πιο καθυστερημένα εισέρχονται στην αγορά εργασίας είναι οι εργαζόμενοι, γι' αυτό και οι συνδρομές στο συνταξιδοτικό μας σύστημα μειώνονται. Αναζητούμε λοιπόν νέε θέσει απασχόληση προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε το συνταξιοδοτικό μα σύστημα και προσπαθούμε να δούμε δουλειέ και για του πιο ηλικιωμένου. Γιατί έχουμε ε, πολλέ φορέ αγορέ εργασία που δημιουργούν διακριτική μεταχείριση ει βάρο των ηλικιωμένων. Θα πρέπει αυτό να το διορθώσουμε και να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης, παρά να δούμε με τεχνικό τρόπο πώς θα αλλάξουμε το σύστημα. Το λόγο θα δώσω τώρα στον κύριο Μίλε από την Ουγγρική Βουλή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι περισσότεροι προλαλήσαντες εμ, προσέγγισαν το πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, το όριο ηλικία η δεξιοδότηση είναι πολύ, χαμηλό από τις, ε, πολύ χαμηλότερο από τις άλλες χώρες. Θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Επίσης, ε, το θέμα της μετανάστευσης είναι διαφορετικό. Έχουμε όλο και μεγαλύτερη έξοδο των νέων από την Ουγγαρία και όλο πιο, όσο πιο ειδικευμένοι νέοι, τόσο περισσότερο έχουν την τάση να αναζητούν ε, θέσεις εργασίας αλλού. Αυτό είναι ένα πλήγμα στην, για τη χώρα μας. Επίσης υπάρχει ε, πρόβλημα και για την κοινωνική δομή, γιατί έχουμε διαρροή ε, εγκεφάλων και διαρροή ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Και οι νέοι που παραμένουν στην Ουγγαρία και αυτοί έχουν πρόβλημα ανέβρεσης δουλειάς. Η δομή λοιπόν του, της αγοράς εργασίας ε, στην Ουγγαρία είναι προβληματική και μια τέτοια φυσικά κοινωνία δεν είναι βιώσιμη. Αυτό σε συνδυασμό με την ε, δημογραφική ε, κατάσταση και την έλλειψη των ανταγωνιστικότητας δημιουργεί μια ζωφερή εικόνα για την ουγγρική κοινωνία και οικονομία. Επίσης εντός της κοινωνίας μεγαλώνουν οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων και ομάδων, κάτι που επιτείνει την κοινωνική ένταση. Είναι πολύ χρήσιμες λοιπόν τέτοιες συναντήσεις μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί μια και συζητάμε και το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, για το 2014 με 2020, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο ποια έμφαση θα δώσουμε. Είμαι μέλος του κόμματος των οικολόγων, γι' αυτό και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δοθεί έμφαση στο περιβάλλον, στην αηφόρο ανάπτυξη, στους τοπικούς πόρους, και στην αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τους νέους και μάλιστα είτε στην περιφέρειά τους είτε στην χώρα τους προκειμένου να μην χρειάζεται να αποδημήσουν. Μία άλλη λύση κατά τη γνώμη μου βρίσκεται στην ενίσχυση της πολιτικής συνοχής και στην καλύτερη κατανομή των κονδυλίων της συνοχής προκειμένου να γεφυρωθούν τα χάσματα και να ανακουφιστεί η κοινωνική πίεση και ένταση που διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση και των γυναικών, ώστε μετά την γέννηση του παιδιού να μπορούν να επανέλθουν και να ανακτήσουν την προηγούμενη θέση εργασίας τους. Σας ευχαριστώ κύριε Μίλε. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Τσίχον και μετά στον κύριο Τσερβίνσκι, τον εισηγητή μας για τα τελικά συμπεράσματα, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο τινά. Γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπε ο εκπρόσωπος ε, της Κυπριακής Βουλής και ο κύριος ε, Αγκούστιν, ο Πολωνός Γερουσιαστής. Ε, ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το περιφερειακό επίπεδο και το εθνικό και σε κάθε ε, επίπεδο να αναλυφθούν δράσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Να μην ξεχάσουμε λοιπόν και την περιφερειακή διάσταση. Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά το εξή. Πολλές φορές μιλούμε για προκλήσεις και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά αποτελέσματα της γύρας πληθυσμού. Αλλά ξεχνούμε μερικές φορές ε, τη θετική πτυχή, τις ευκαιρίες που μας δίνει ε, αυτό το φαινόμενο. Γιατί ε, ο γυράσκον πληθυσμό που έχει ιδιαίτερε ανάγκες μπορεί και αυτός να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη με την ε, δημιουργία νέων αγαθών και υπηρεσιών ή με την ενίσχυση υπηρεσιών που ικανοποιούν ιδιαίτερα τις ανάγκες των ηλικιωμένων. Ε, και η ανάπτυξη τέτοιων αγαθών και υπηρεσιών μπορεί να συμβάλλει στην ε, δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση όχι μόνο για ηλικιωμένους αλλά και για νέους. Και κάτι άλλο, οι ηλικιωμένοι που ζουν όλο και περισσότερο είναι και ε, σωματικά αλλά και ψυχικά υγιείς. Αυτό το δυναμικό θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Πολύ συχνά το ξεχνάμε αυτό και το εξετάζουμε μόνο τη δημογραφία υπό το αρνητικό πρίσμα του προβλήματος. Αυτά λοιπόν ως προς το πρώτο πάνελ και θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο στον Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για να σχολιάσει αυτά που ακούσαμε και μετά στον εισηγητή μας. Ευχαριστώ. Thank ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα αρκετές παρατηρήσεις οι οποίες θα πρέπει να τύχουν απάντησης. Καταρχάς να πω ότι η συζήτηση ήταν πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα. Έχω εδώ πέντε ή έξι στοιχεία τα οποία νομίζω όμως ότι θέλουν διευκρινήσεων. Πρώτον, ένας από τους συναδέλφους από το Ηνωμένο Βασίλειο τόνισε ότι υπάρχει μάλλον ε, μία αντίφαση ανάμεσα στην υψηλή ανεργία από τη μία και την ανάγκη αύξησης του ηλικία συνταξιοδότησης. Λέτε στην ουσία βέβαια ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και ποιος θα τις δημιουργήσει. Βέβαια η τεχνική απάντηση υπάρχει. Εμείς κάναμε κάποιες προβολές και στο παρόν επίπεδο και με το παρόν ποσοστό απασχολησιμότητας και με τις προβλεπτές δημογραφικές εξελίξεις η αντίφαση αυτή θα χαθεί από τον ορίζοντα το 2020 με 25 σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να εξαφανιστεί αυτή η ανισορροπία, όχι στο σύνολο, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, σε πάρα πολλές περιοχές. Η κρίση ίσως να έχει αναβάλει βέβαια και καθυστερήσει αυτή την αποκατάσταση κατά μια πενταετία περίπου, αλλά δημογραφική λύση προβλέπεται. Εδώ υπάρχει μια προφανής όμως αντίφαση. Αν είσαι ένας άνεργος νέος, θα σου ζητούσα και μπορείς να ανταποκριθείς αυτό καλύτερα από μένα, τι μπορείς να κάνεις για να γίνεις απασχολήσιμος. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την εκπαίδευση όμως των νέων. Ε, υπάρχει έλλειμμα στην εκπαίδευση, υπάρχει έλλειμμα στην τεχνική κατάρτισή τους, υπάρχει έλλειμμα στην προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας. Μήπως απαιτούνται επενδύσεις σε αυτό το πρόωρο στάδιο, σε αυτή την πρόωρη φάση σε μια κοινωνία η οποία από ό,τι φαίνεται μεγαλώνει τα παιδιά της με όλο και περισσότερες δυσκολίες και τα εκπαιδεύει με όλο και περισσότερες δυσκολίες. Η δημοσιονομική πειθαρχία και οι περικοπές κατά από τα μέτρα τα περιοριστικά έχουν λάθος στόχο. Χτυπούν τα συστήματα εκπαίδευσης και βλέπουμε ε, ποιες είναι οι αρχές των αρνητικών επιπτώσεων σε σχέση με την απασχολησιμότητα σαν παράδειγμα των νέων. Σημειώνω ένα άλλο θέμα που τέθηκε, ότι δεν μπορούμε εμείς να αντέξουμε πλέον το κράτος προνοίας. Ποιος το είπε αυτό, ποιος σας το λέει αυτό, γιατί το αναδιανεμητικό σύστημα δεν παρεμποδίζει την ανάπτυξη, η ζήτηση δεν θα πρέπει να μειωθεί μόνο και μόνο λόγω της ανακατανομής του εισοδήματος, αυτό είναι μύθος. Ακόμα και αν δείτε το σύνολο των οικονομιών των ευρωπαϊκών θα δείτε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην αναδιανομή και ταυτόχρονα αυτές οι τεράστιες αλλαγές δεν αντικατοπτρίζουν σε καμία περίπτωση τις οικονομικές επιδόσεις των ίδιων χωρών. Αν κάποιος λέει ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε το κράτος προνοίας εννοεί ότι υπό το παρόν καθεστώς καλύψεων και φορολογίας πράγματι λογιστικά έχουμε πρόβλημα. Αλλά γιατί είναι δεδομένα τα ποσοστά αυτά των εισφορών σαν παράδειγμα των συμμετεχόντων στο σύστημα. Γιατί θα πρέπει διαγενειακά να καθορίσουμε το επίπεδο φορολογίας γιατί υπάρχουν και οι διαφορές ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Γερμανία και στη Σουηδία. Γιατί να το πω καλύτερα, στη Σουηδία το κόστος των συνεισφορών είναι κατά 13% υψηλότερο από ό,τι στη Γερμανία σαν παράδειγμα. Λοιπόν ήταν ένα παράδειγμα. Το θέμα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Είναι θέμα της πολιτικής βούλησης. Δεν θέλουν να υπάρξει μεγαλύτερη αναδιανομή από ό,τι το παρόν σύστημα. Αλλά δεν είναι τίποτα το δεδομένο αυτό, δεν είναι κάτι το θέσφατο, μπορεί να αλλάξει. Το μήνυμα ποιο είναι. Υπάρχουν περιοχές στην Ευρώπη όπου πρέπει να αυξηθεί η φορολογία. Και μπορεί να αυξηθεί η φορολογία. Και όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο είναι κάτι το οποίο προφανώς ε, ε, θα πρέπει να οδηγήσει στην αναζήτηση μιας διαφορετικής λύσης. Αλλά το να πούμε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, να αυξήσουμε την φορολογία και να αυξήσουμε τις ε, συνεισφορές, αυτό είναι μύθος. Προφανώς 100% δεν μπορούμε να τα αυξήσουμε, αλλά υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούν να αντέξουν την αύξηση των συνεισφορών και των φόρων. Μπορούμε λοιπόν να βρούμε πολιτικές λύσεις εφόσον έχουμε μια κοινή αγορά αγαθών, υπηρεσιών, έχουμε ελεύθερη διακίνηση προσώπων και θα πρέπει να παραμείνει το καθεστώς αυτό, τότε γιατί να μην, να μην βρεθούν ευρωπαϊκές λύσεις. Αυτή τη στιγμή το διακανονιστικό σύστημα δεν ρυθμίζεται μέσω αμυγός εθνικών μέτρων και αυτό θα πρέπει να αλλάξει θα πρέπει να υπάρξει ανάγκη σε εκεί όπου απαιτείται. Υπάρχει κάτι το οποίο αγνοούμε μερικές φορές. Συμφωνώ με αυτούς οι οποίοι το είπαν, ότι σε ορισμένες περιοχές, στο Ηνωμένο Βασίλειο σαν παράδειγμα, υπάρχει υπερβολική πυκνότητα πληθυσμού σε σχέση με την απασχόληση. Από την άλλη όμως, αν θέλουμε τα πράγματα να προχωρήσουν, θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις απαιτούμενες επενδύσεις. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές που θα οδηγήσουν τις επενδύσεις. Όταν θέλουμε να μην φεύγει ο κόσμος από περιοχές τις οποίες ε, αυτή τη στιγμή εγκαταλείπει, τότε θα πρέπει να αντιστρέψουμε τις χρηματοπιστωτικές ε, ε, ροές αν τα χρήματα έρχονται από το α στο β συστηματικά και μακροπρόθεσμα, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και θα πρέπει να αλλάξει. Τότε μόνο δεν θα φεύγουν οι δραστήριοι επαγγελματικά από συγκεκριμένες οικονομίες για να πηγαίνουν σε άλλες. Δεν υπάρχει άλλη λύση προς το παρόν εκεί. Και ποτέ δεν είπα εγώ ότι η μετανάστευση είναι η μόνη λύση. Όχι, τα μοντέλα τα οποία διατυπώσαμε, τα οποία προτείναμε, λένε ότι αν είναι να απολογίσουμε μέχρι το 2015, τότε κάθε χρόνο ή στα πλαίσια της πενταετούς, εμπασπέντος χοντρικά περίοδου, μπορούμε να ορίσουμε τον αριθμό των μεταναστών έτσι ώστε να αντισταθμίσουμε ε, τα δημογραφικά στοιχεία. Αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα γιατί οι μετανάστες συνήθως ε, υιοθετούν το αναπαραγωγικό πρότυπο της κοινωνίας που τους φιλοξενεί. Οπότε θα εξακολουθήσουμε να έχουμε προβλήματα και τις επόμενες δεκαετίες ε, θα έχουμε προβλήματα διατήρησης του καθεστώτος έτσι όπως ισχύει σήμερα. Πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε από τη μία υψηλότερα ποσοστά απασχολησιμότητας και υψηλότερα ποσοστά μετανάστευσης. Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στα παιδιά και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε την αγορά εργασίας με τρόπο ο οποίος σίγουρα σήμερα δεν είναι εύκολος. Και δεν είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά λέμε ότι αν πράγματι μπορούμε να κρατήσουμε έναν χαμηλό σταθερό ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη, αυτό θα βοηθήσει έτσι ώστε οι διάφορες περιοχές της Ευρώπης να μπορέσουν να έλθουν πιο κοντά. Και οι διαφορές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των περιφερειών των περιοχών θα πρέπει να είναι ανεκτού τύπου και θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα μετακινήσεων πληθυσμών προσωρινά έστω για την κάλυψη των τοπικών αναγκών. Θυμάστε ότι στη δεκαετία του 90 υπήρχαν κάποιες μεταναστευτικές ροές, αλλά τώρα μετά από τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν σε ορισμένες χώρες, οι ίδιοι άνθρωποι συνεχίζουν κατά κάποιο τρόπο τη μετανάστευσή τους προς άλλες περιοχές. Ένα άλλο θέμα, τελευταίο θέμα. Απαιτούνται δημόσιες επενδύσεις. Δεν μπορώ εγώ να είμαι πεπισμένος ότι η αγορά θα επενδύσει από μόνη της και θα βρει μόνη της λύση για να ε, αντιμετωπιστούν τα δημογραφικά προβλήματα σε 20-30 χρόνια. Όχι, αυτό δεν θα το κάνει η αγορά. Πρέπει το κράτος να επενδύσει στην εκπαίδευση, πρέπει να επενδύσει στην διαβίου κατάρτιση, αυτό θα κοστίσει φυσικά και αν έχετε κάποιον με 40 χρόνια επαγγελματική σταδιοδρομία και ξαφνικά θα πρέπει να τον εκπαιδεύσετε για 4 χρόνια, προφανώς αυτό θα αυξήσει πάρα πολύ το κόστος εργασίας και το κόστος των επενδύσεων, των δημοσίων. Αυτό θα το κάνει όμως το κράτος, δεν θα το κάνει η αγορά. Και οι φόροι που πληρώνουμε σήμερα θα πρέπει να επενδύονται έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε σε 20-30 χρόνια. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της απασχόλησης σε 10, 20, 30 χρόνια απαιτούνται μακροπρόθεσμες λύσεις, απαιτείται επένδυση θα έλεγα εκ των προτέρων και αυτή η εκ των προτέρων επενδυτική προσπάθεια πρέπει να γίνει ανεκτή από τον πληθυσμό γιατί δεν το καταλαβαίνει εύκολα ο γενικός πληθυσμός αυτό. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε όλο τον κόσμο. Τα μέτρα που παίρνονται είναι περιοριστικά και αντιπαραγωγικά. Το θέμα είναι ότι απαιτούνται μακροπρόθεσμες επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσίχων γιατί αναφερθήκατε σε ορισμένα από τα θέματα και τη συζήτηση. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γιαντών από την Εσθονική Βουλή και μετά στον εισηγητή μας τον κύριο Τσερβίνσκι για τα τελικά σχόλια. Σας ευχαριστώ. Είναι πραγματικά δύσκολο να παρέμβει κανείς μετά τον προλαλήσαντα. Αλλά θα ήθελα να τονίσω κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, προέρχομαι από μια μεθοριακή περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέμε ότι Όσο πλούσιος και να είναι κανείς ή όσο φτωχός και να είναι κανείς ε, δεν ικανοποιείται με αυτή την κατάσταση πραγμάτων και το πώς ε, διαμορφώνονται τα πράγματα. Και το βλέπουμε και αυτό σήμερα. Ο εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου είπε δεν υπάρχει πρόβλημα με το ποσοστό γεννητικότητας διότι καλύπτεται αυτό ε, από την οι ανάγκες καλύπτονται από το ποσοστό γεννητικότητας. Όμως και σε σχέση με τη μετακίνηση από τη χώρα μας ε, εργαζομένων προς τις ε, άλλες χώρες, ε, πιο προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας ικανοποιεί. Όταν κάνουμε λόγο για την χρήση μεταναστών σε σχέση με την αγορά εργασίας, υπάρχουν διαφορές εδώ σε αυτό, το, σε αυτό το τομέα. Ένα άλλο πράγμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι η ηλικία συνταξιοδότησης. Όπως ανέφερε και ο Ούγγρος συνάδελφος, το προσδόκιμο ζωής είναι χαμηλότερο στην Εσθονία ή στην Ουγγαρία από ότι ε, το προσδόκιμο ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στη Γερμανία. Και η υγεία μας είναι επιδεινωμένη, βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα. Στην Εστονία δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται ε, πολλοί επειδή ασθενούν. Ε, έχουν, είναι ε, ηλικιωμένοι, ασθενούν, πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις διαφορετικές αυτές περιπτώσεις. Όλα αυτά τα προβλήματα δεν μπορούν ε, με πανάκια να επιληθούν. Με αισιοδοξία αντιμετωπίζω τα πράγματα και ελπίζω ότι οι Ευρωπαϊκέ χώρε θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν αυτά τα προβλήματα από κοινού, ενωμένε. Βλέπουμε όμω ότι οι περισσότερε χώρε αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ακολουθήσουν τα ξεχωριστά δικά του συμφέροντα. Προσπαθώ με πνεύμα επικοδομητικό να αντιμετωπίσω τα πράγματα. Κάποιο αναφέρθηκε στην αργυρή οικονομία, silver economy. Θα ήθελα να ακούσω από του συναδέλφου τι συμβαίνει να μας δώσουν καλά παραδείγματα, πρότυπα, πώς θα μπορούσαν ε, οι ηλικιωμένοι ε, που έχουν ασπρίσει τα μαλλιά τους Silver Economy XU, πώς θα μπορούσαν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Πρέπει να δούμε ποια συμπεράσματα μπορούμε να συναγάγουμε. Τα γεράματα δεν μπορεί κανείς να τα θεραπεύσει και υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου οι ηλικιωμένοι θα μπορούσαν να είναι παραγωγικοί και να εργάζονται. Στην Εστονία το επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και παιδείας είναι υψηλό. Οι, εκπαιδε... μορφωμένοι που μιλάνε και δύο-τρεις γλώσσες μπορούν μέχρι και τα προχωρημένα γερατιά τους να απασχοληθούν και να εργάζονται. Αν δεν έχουν αυτή την παιδεία και εκπαίδευση δεν μπορούν να εργάζονται. Θέλω να μας πείτε ποια είναι τα καλύτερα παραδείγματα λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους και των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συμμετοχή τους στη συζήτηση και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Σερβίνσκι, για να μας κάνει μια ανακεφαλαίωση και να υποβάλει τα τελικά συμπεράσματα. Κύριε Τζέι Τσερβίνσκι, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη ευρωβουλευτά και βουλευτέ, οι οργανωτές, οι διοργανωτές μου ζήτησαν να αντλήσω κάποια συμπεράσματα ε, και να κάνω κάποια ανακεφαλαίωση της συζήτησης. Φυσικά είμαι υποχρεωμένος να κρατήσω το την ίδια κατεύθυνση με αυτή που σας παρουσίασα στην αρχή. Δηλαδή, ε, να προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση ήταν υπάρχει πραγματική απειλή αν δεν ε, αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Όλοι όσοι λάβατε το λόγο υπογραμμίσατε το πρόβλημα και ε, επισημάνατε κάποιους τρόπους για την επίλυση. Το θέμα είναι, θα πρέπει ήδη από τώρα να αναλάβουμε κάποιες προσπάθειες γιατί είναι πραγματική απειλή της όξης της κρίσης και της επιδήλωσης του προβλήματος. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, ποιος θα πρέπει να αναλάβει αυτές τις δράσεις αφού κρίθη απαραίτητο να αναλυφθούν. Ήταν πολύ ευχάριστο που πολλοί είπαν και θα έλεγα όλοι. Κανένα δεν επέριψε το πρόβλημα στον άλλον, εκτό και αν κάποιο το έκανε και δεν το αντιλήφθηκαν εγώ. Νομίζω ότι όλοι αναγνώρισαν ότι είναι απαραίτητη η ανάληψη δράσεων σε εθνικό επίπεδο, αλλά ε, είναι απαραίτητο και ο συντονισμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό, αυτό το συμπέρασμα μπορεί να γίνει δεκτό από όλους και αν το δεχτούμε πραγματικά θα έχουμε, ε, ένα, θα έχουμε πραγματοποιήσει ένα ποιοτικό άλμα πολύ σημαντικό στην κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος. Ακούσαμε ότι είναι ιδιαίτερα δρυμή το πρόβλημα της ανεργίας. Θα μπορούσαμε να ομαδοποιήσουμε κάπως τα προβλήματα και νομίζω ότι ένας τρόπος, ε, θεμελιώδης τρόπος ε, για να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα είναι η οικονομική ανάπτυξη. Με την οικονομική ανάπτυξη δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Και η οικονομική ανάπτυξη ε, περιορίζει και τον αριθμό των ανέργων. Επίσης, η οικονομική ανάπτυξη δίνει κίνητρα και θαρρύνει και τους νέους ε, να εισέλθουν στην αγορά εργασία. Δεν θα ήθελα να αναφέρω τους όρου και τι προποθέσει της οικονομική ανάπτυξη. αλλά νομίζω ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι δυνατή και πιθανή μόνο όταν και τα δημοσιονομικά ενό κράτου βρίσκονται σε υγιή και σταθερή κατάσταση. Και γι' αυτό θα, θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση προ τα κράτη-μέλη να προσέξουν ιδιαίτερα αυτές τις προϋποθέσεις για την υγιή δημοσιονομική διαχείριση και τα σταθερά οικονομικά. Αυτό φυσικά θα πρέπει να γίνει και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φυσικά υπάρχουν πολλές διαφορές. Ε, άλλες συνθήκες επικρατούν στη Σουηδία και άλλες στο Ηνωμένο Βασίλειο, άλλες ε, στην Εστονία και άλλες ε, στην Ουγγαρία. Θα πρέπει πάντως όλοι να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιαίτερες ηθίκες σε κάθε χώρα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό συμπέρασμα, μια και έχουμε ένα κοινό μακροπρόθεσμο στόχο. Ο κοινός μας στόχος είναι η σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας και το μέλημα για να εξασφαλίσουμε ε, βιώσιμο μέλλον και στους ε, και στις επερχόμενες γενιές. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε συντονισμό των πολιτικών, όχι μόνο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα τελευταίο ζήτημα το οποίο ανέκυψε και θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε αυτό. Ίσως ε, δεν το λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη κάποιοι εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες, ε, ε, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Η επικοινωνία με τους πολίτες, οι επαφές με τους συμπολίτε μας, γιατί οι πληροφορίες είναι σημαντικές όχι μόνο μεταξύ μας και η ενημέρωση, είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι πολίτες, ε, να ξέρει η κοινωνία ποιοι, ποιοι είναι οι όροι και με ποιες προϋποθέσεις θα υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Και όπως είπατε και οι περισσότεροι από εσά, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι χωρίς επικοινωνία με τους συμπολίτε, χωρίς ενημέρωση του κάθε πολίτη για την κατάσταση, πολύ δύσκολο θα είναι από κοινού να υλοποιήσουμε τον κοινό μα στόχο. Χρειαζόμαστε αυτή την σωστή ενημέρωση και επαφή με του πολίτε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τζέι Τσερβίνσκι, βουλευτή της Πολωνικής Βουλής, του ΣΕΙΜ, που ήταν ο συγητής μα, αλλά να ευχαριστήσω και όλους όσους έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Φάνηκε από τη συζήτηση ότι ήταν πολύ σημαντικό το θέμα, αλλά καταφέραμε να ολοκληρώσουμε εγκαίρως τη συζήτηση του πρώτου πάνελ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω τη σκητάλη στο δεύτερο πάνελ και στους δύο συμπρόεδρους, την κυρία ε, Ντανούτα Χίμπνερ που είναι εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, στον κύριο ε, Άντζε Γκαουαζεύσκη που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων στην Πολωνική, από την Πολωνική Βουλή. Ευχαριστώ.

Πρωτού ξεκινήσουμε με το δεύτερο πάνελ, αν μου επιτρέπετε. Θα ζητήσω από τον κύριο Μπουσέβιτς να παρουσιάσει, να κάνει αυτή την εισαγωγή, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να χαιρετήσω την κυρία Κρέλη, συγκεκριμένα Ευρωβουλευτήνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κυρία Ντανούτα Χύμπνερ, Ευρωβουλευτήνα, που την χαιρέτησε προηγούμενα ο προλαλής σας, αγορητής ο κύριος Γκαζεύσκη. θα είναι και κοντά μας, ο κύριος Γκαζεύσκη. Η κυρία Κρέλη έχει πέντε λεπτά για να προετοιμαστεί αυτή η συζήτηση και να κάνει την εισαγωγή της. Παρακαλώ κυρία Κρέερ. Χωρίς μικρόφωνο. Με μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Χίμνερ, αγαπητοί συνάδελφοι, για μένα είναι κάτι καινούριο, καινοτόμο να βρίσκομαι εδώ μπροστά Κανονικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλάμε από το έντρανό μα, από τη θέση μα. Ευχαρίστω όμω να παρέμβω με αυτόν τον τρόπο, από αυτή τη θέση εδώ. Ελπίζω ότι όπω πάντα η διερμηνία θα είναι εξαιρετική. Λοιπόν, ο συνάδελφο Φανίστερ Ρόι και εγώ είμαστε συνεισηγητέ και οι δύο για τον γενικό κανονισμό και γνωρίζετε ότι αρχές Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νομοθετικό πακέτο μέτρων το παρουσίασε για τη μελλοντική πολιτική συνοχή και από τότε εργαζόμαστε εντατικά σε αυτό το πεδίο και έχουμε και ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο εγκρίναμε και ελπίζουμε ότι κατά τα τέλη του 2012 πραγματικά θα έχουμε συμφωνήσει για τις θέσεις μας για ένα κοινό νομοθετικό πακέτο μέτρων για την μελλοντική πολιτική συνοχή. Αυτό εξαρτάται όμως επίσης από το ότι αν η μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση θα έχει συμφωνηθεί και θα έχει εγκριθεί εντωμεταξύ, διότι χωρίς κονδύλια δεν μπορεί κανείς να εγκρίνει νομοθετικό έργο. Ελπίζω ότι όλοι θα καταβάλουν προσπάθειες και ότι το Συμβούλιο των Υπουργών θα έχει και εκείνο συμφέρον, όπως και το Ευρωκοινοβούλιο, το δυνατόν νωρίτερα να ολοκληρώσουν και από το Συμβούλιο με τις προκατακτικές εργασίες για να εγκριθούν όλα αυτά. Πρώτον και κύριον πρέπει να πω ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα ότι υπέβαλε αυτές τις προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτές οι προτάσεις καταδεικνύουν ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και πρέπει να αντιμετωπιστούν και μετά το 2014 στο πεδίο της συνοχής. Και είναι ιδιαίτερα θετικό ίσως το ότι πολλές προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήδη, ήδη εντάχθηκαν και από πλευρά της έκθεσης Πίπερ στην έκθεση συνοχής που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι αντανακλώνται στο νομοθετικό πακέτο μέτρων, στη δέσμη μέτρων του νομοθετικού αυτού ε, προγράμματος. Και είναι καλό το ότι έχει δεχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προτάσεις ότι όλες οι περιφέρειες και περιοχές της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης πρέπει να συμμετέχουν και να υποφεληθούν από την πολιτική συνοχή. Γνωρίζουμε ότι υπήρχαν πολύ διαφορετικές θέσεις και τοποθετήσεις και πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό μήνυμα ακριβώς σε αυτό το πεδίο στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιοχές και επαρχίες μας να γνωρίζουν ότι θα τύχουν τις αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπαινος τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση στο Γενικό Κανονισμό ότι για πρώτη φορά όλα τα ταμεία συμμετέχουν. Όχι μόνο το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης και το Κοινωνικό Ταμείο, αλλά και το Ταμείο Ανάπτυξης Υπέθρου και το Ταμείο για την Αλληλεία. Και έτσι είναι δυνατόν μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο μια απλουστευμένη διαδικασία για όλα αυτά τα ταμεία να εγκριθεί και να λειτουργήσει. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε βελτιωμένο συντονισμό μεταξύ των ταμείων και των δράσεων των ταμείων που θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων. Η νέα πολιτική συνοχής λοιπόν σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεσμεύεται με την πολιτική για την συνοχή, με την ενίσχυση της ε, περιφερειακής συνεργασίας και την διαμεθοριακή, διασυνοριακή συνεργασία. Το πιο σημαντικό μέσο όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής, της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 καθίσταται σαφές από τις προτάσεις που έχουμε μπροστά μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιο είναι αυτό το πλαίσιο. Έχουμε κάποια σημεία λοιπόν που πρέπει να τύχουν ιδιαίτερη συζήτηση και προσοχή. Και ελπίζω ότι και κατά τη διάρκεια του σημερινού απογεύματο θα γίνει αυτό. Πρέπει να δούμε σε ποια σημεία πρέπει να προβληματιστούμε πιο έντονα. Να δούμε τι πρέπει να διαμορφωθεί και τι πρέπει να εξειδικευθεί με καλύτερο τρόπο για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Κάποια σημεία θέλω να αναφέρω, διότι πιστεύω ότι στη συζήτηση στη συνέχεια θα έχουν τη μεγάλη σπουδαιότητα αυτά. Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο λοιπόν να έχουμε μια ισορροπία που πρέπει να εξεύρουμε μεταξύ αφενός της κατεύθυνσης των κατευθύνσεων για τη στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020 και των συμφερόντων των περιοχών και περιφερειών ώστε με πιο αποτελεσματικό τρόπο να θεσπίσουμε προτεραιότητες για τις περιφέρειές μας, ανάλογα με τις πραγματικές τους ανάγκες πάντα. Πιστεύω ότι με τις εταιρικές ε, συμφωνίες και ε, ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτές τις περιφέρειες, πρέπει να μπορέσουμε να δράσουμε με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανάλογα με τις ειδικέ ανάγκες που έχουν αυτές οι περιφέρειες. Διαπιστώνουμε ότι και πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ΑΕΠ χρησιμοποιεί ως βάση για την υποστήριξη και συνδρομή σε σχέση με αυτές τις περιφέρειες. Έχουμε δύο κατηγορίες τις λιγότερο ανεπτυγμένες ε, ή τις λίγο ανεπτυγμένες περιφέρειες, στόχος 1, που ε, βρίσκονται κάτω από το 75% ή προσεγγίζουν το 75% του ΑΕΠ και οι περαιτέρω ανεπτυγμένες περιοχές ε, που βρίσκονται πάνω από αυτό το ποσοστό. Τώρα έχει υποβάλει μια νέα πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το Κοινοβούλιο πλειοψηφικά υποστηρίζει, δηλαδή μια νέα ενδιάμεση κατηγορία, μια ενδιάμεση ομάδα περιφερειών ε, να θεσπιστεί δεδομένων πολλών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες ενδιάμεσες περιοχές μεταξύ 75% και 90% του ΑΕΠ, του μέσου όρου ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου με ιδιαίτερο τρόπο θα υποστηρίζονται στον ευάλωτο χαρακτήρα τους αυτές οι περιφέρειες. Για παράδειγμα, έχουμε και περιφέρειες που βρίσκονται στο 180 περίπου της 100 του ΑΕΠ και πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις διαφορές που υπάρχουν εναντί άλλων περιφερειών. Αν γίνει αυτό, τότε θα έχουμε μια καλή προϋπόθεση για την μελλοντική συνεργασία και θετικά αποτελέσματα για την πολιτική συνοχή. Ένα ουσιαστικό θέμα στο οποίο δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα για τα παράπονα που εκφράζονται από τις περιφέρειες ότι υπάρχουν η γραφειοκρατική επιβάρυνση, γραφειοκρατική ε, επιβράδυνση, όχι μόνο επιβάρυνση αλλά και επιβάρυνση λόγω της γραφειοκρατίας εξετάζουμε τις δυνατότητες απλούστευσης σε σχέση με τα μέτρα που έχουν προταθεί για να δούμε μήπως δημιουργούνται πρόσθετες δυσκολίες. Θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε το θέμα των όρων και προϋποθέσεων. Πώς θα την χάνουν υποστήριξη σε αυτές οι περιφέρειες. Εδώ υπάρχει ανάγκη διαβούλευσης και συζήτησης και ελπίζω ότι και από εσάς θα υπάρξουν προτάσεις και απόψεις που θα εκφραστούν για να βελτιωθεί αυτό το πλαίσιο. Και στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να συζητήσουμε για μια ενισχυμένη παράμετρο για τα αστικά κέντρα, που δεν θα ξεχνά όμως και το χώρο της υπαίθρου με κανένα τρόπο. Θα πρέπει παράλληλα να εξετάσουμε αυτές τις ανάγκες οι πόλεις που πραγματικά τα αστικά κέντρα που σχεδόν 80% συλλέγουν ε, του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν σε αυτές τις πόλεις, η πολιτική συνοχή θα πρέπει να αναπτυχθεί με ιδιαίτερα αηφόρο τρόπο ως προς αυτές τις παραμέτρους για να υποστηρίξουμε τους, τις ανάγκες των πολιτών μας. Όπως γνωρίζετε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνδέεται και με μια δημοσιονομική πρόταση. Σύμφωνα με την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 376 δισεκατομμύρια ευρώ θα ε, διατεθούν για την, ε, το μέσο διευκόλυνσης για να μπορέσει να υποστηριχθεί αυτή η προσπάθεια. Πρέπει να διασφαλιστεί από το Συμβούλιο ότι θα διατεθούν αυτά τα χρήματα. Πρέπει σίγουρα να συζητήσουμε πώς το Connecting Europe, η διαδικτύωση της Ευρώπης, ε, η συνένωση της Ευρώπης μέσα από αυτό το εγχείρημα θα μπορέσει να καλυφθεί. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κρέλ. Πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση, θα ήθελα να σας πω ότι όσοι θέλουν το λόγο θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο μοιράστηκε σε όλες τις αντιπροσωπείες. Εμείς θα προετοιμάσουμε έναν κατάλογο για να ορίσουμε τους ομιλητές. Δύο κοινοβούλια. Εθνικά κοινοβούλια, δύο εθνικά κοινοβούλια, ένας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δύο λεπτά ο καθένας. Θα έχετε το χρονόμετρο μπροστά σας. Και η Προεδρία θα αποφασίσει αν θα ξεκινήσει τη διαδικασία της μπλε κάρτας. Παρακαλώ, λοιπόν, εγγραφείτε για τη συζήτηση και ξεκινάει η συζήτηση. Από τη Λιθουανία, ο κύριος Κορπουέσας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. νέα Πολιτική συνοχής είναι μία από τις ε, κύριες ε, ευρωπαϊκές πολιτικές που θα συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα. Θα δίνει πρόσθετη αξία, θα δίνει τη δυνατότητα της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής και της ε, περιφερειακής ανάπτυξης. Στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για το 2014 έως το 2020 η πολιτική συνοχής θα διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής συνολικά για την Ευρώπη του 2020. Είναι λοιπόν για αυτούς τους λόγους σημαντικό αυτή η πολιτική να είναι ενδυναμωμένη, να είναι ισχυρή και αποτελεσματική. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το νόημα της ε, πολιτικής συνοχής είναι να μειωθεί βελτιωθούν οι διαφορές στα επίπεδα περιφερικής ανάπτυξης μεταξύ των χωρών μελών μας. Και η προτεραιότητα πρέπει πάντα να έγκυται <clears throat> στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει ιδιαίτερα να υποστηρίζονται. Τώρα, όσον αφορά τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό που μεριμνούμε και ε, μας κάνει να ανησυχούμε είναι να καλύψουμε τις ε, προϋποθέσεις όσον αφορά το ποσοστό ΑΕΠΑ. Τι σημαίνει όμως αυτό, ότι η υποστήριξη για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές θα μειωνόταν από το 81% στο 68% περίπου. Και για αυτούς τους λόγους ε, οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και περιοχές της Ένωσης θα βρίσκουν ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να καλύψουν το χάσμα που τις χωρίζει από τις πιο προηγμένες περιφέρειες. Οι αλλαγές λοιπόν όσον αφορά την, ε, τους πυλώνες στήριξης θα πλήξουν ε, ιδιαίτερα τις περιοχές εκείνες που το ΑΕΠ τους επλήγει ακόμα περισσότερο και μειώθηκε, συρρυκνώθηκε λόγω της κρίσης. Και αυτό σίγουρα θα επιβραδύνει τη διαδικασία μείωσης των χασμάτων και κάλυψης των κενών μεταξύ λιγότερων επιμένων περιοχών και περισσότερων προηγμένων περιοχών θα έπρεπε να υιοθετηθεί μια δυνατότητα επιτάχυνσης, επιταχυμένης δυνατότητας προσέγγισης των στόχων. Αν δεν ε, ακολουθήσουμε μια τέτοια πολιτική θα υπονομευθούν οι στόχοι της στρατηγικής του 2020. Θα θέλαμε επίσης να συζητήσουμε και το ελάχιστο επίπεδο, τα ελάχιστα επίπεδα τα οποία θα πρέπει να θεσπιστούν και για τις ελάχιστες διαστάσεις ή ελάχιστες αναλογίες ή ποσοστά που θα θεσπιστούν όσον αφορά τα κονδύλια του προϋπολογισμού που θα δίνονται από το Ταμείο Συνοχής ε, και το, ταμείο, το Κοινωνικό Ταμείο για την επίτευξη αυτών των στόχων. Δέκα δις ε, αναφέρονται από πλευρά του Ταμείου Συνοχής ε, για το Ευρωπαϊκό Μέσο Υποδομών. Οι αρχές μεταφοράς αυτών των κονδυλίων είναι ασαφείς ακόμα. Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι ειδικοί όροι ε, για την χορήγηση αυτών των κονδυλίων και την λειτουργία των προγραμμάτων. Εν τέλει, θέλω να αναφέρω κάποιες ιδέες που θέλουμε να υποστηρίξουμε από πλευράς μας. Εμείς υποστηρίζουμε από πλευράς μας την ιδέα ότι θα πρέπει να θεσπιστεί ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο που θα εμπλαισιώνει και θα εντάσσει και τα πέντε ευρωπαϊκά ταμεία που λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε μεγαλύτερη διασύνδεση και αποτελεσματικότητα δράσεων. Έχουμε και την ανάγκη εξ άντε όρων, εκ προημίου υλοποίηση ε, δηλαδή ε, συγκεκριμένων όρων όσον αφορά και τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Έχουμε κάποιες ανησυχίες ε, πρέπει να πω όσον αφορά το σχέδιο, τα σχέδια εγγράφων που δεν πάνε αρκετά μακριά ώστε να ελαχιστοποιηθεί το γραφειοκρατικό βάρος που επομίζονται τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει και η διοικητική επιβάρηση, το διοικητικό βάρος να απλουστευτεί και να μειωθεί. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και ελπίζω, την, ε, εκφράζω την ελπίδα ότι αυτές οι προτάσεις θα τύχουν ε, προσοχής και συνέχεια. ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Λενέ της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Ο κύριος Λενέ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτό το πάνελ για την πολιτική της κοινωνικής συνοχής σε περιφερειακό επίπεδο να σας αναφέρω μερικά πράγματα τα οποία ανησυχούν ιδιαίτερα τους ε, Γάλλους. Αφορά στις εδαφικές ανισότητες ε, για την πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες. Ξέρετε ότι ο πληθυσμός γερνάει και χρειάζεται να έχουμε θεραπείες ε, και φροντίδες στο ύψος των προσδοκιών των πολίτων. Σήμερα οι στατιστικές του Υπουργείου Υγείας ε, της Γαλλίας προβλέπουν ότι θα μειωθούν οι υπηρεσίες αυτές κατά 10% στα επόμενα 15 χρόνια. Και το 2020 το επίπεδο παροχής υπηρεσιών θα είναι αντίστοιχο εκείνου του 1980. Βλέποντας δε και πόσοι φοιτητές γράφονται σήμερα στη ιατρική, η τάση επιβεβαιώνεται. Πρέπει να δούμε επίσης πώς γίνεται ο καταμερισμός στην επικράτεια. Βλέπουμε μεγάλες γεωγραφικές ανισότητες και έχουμε πραγματικά ιατρικές ερήμους σε ορισμένες περιοχές. Πρόκειται για μια πρόκληση που θα πρέπει να αναλάβουμε για να μπορέσουν να την χάνουν ιατρικών υπηρεσιών όλοι οι πολίτες. Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί έχουν έναν διπλό προς ανατολισμό, έναν μηχανισμό, όπως επίσης και οικονομικά κίνητρα, ούτως ώστε οι φοιτητέ να επιλέγουν ως προορισμό τους ε, ε, απομακρυσμένες περιοχές ή νησιά. Και κίνητρα επίσης ε, στα παραγιατρικά επαγγέλματα για να μπορούν να επιλέγουν δύσκολες περιοχές. Βλέπουμε εμείς ε, πάντως και σήμερα στη Γαλλία ανησυχητικές διαφορές σε αυτό το επίπεδο παροχής υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο και πιστεύω ότι αυτή η πλευρά θα έπρεπε, αυτή η πτυχή θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη στην πολιτική κοινωνική συνοχή για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάμπερτ Βαν Νίστερ Ρόι, Ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ, με βλέπετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μαζί με τη συνάδελφο την κυρία Κρέλ προσπαθήσαμε να σταθούμε στα πιο σημαντικά σημεία σε αυτή τη φάση των συζητήσεων. Απαιτούμε input περισσότερο από τα εθνικά κοινοβούλια. Μιλάμε για την κοινωνική συνοχή σαν παράδειγμα. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το κοινωνικό ταμείο. Το ε, κοινωνικό ταμείο εξακολουθεί να λειτουργεί. Παρ' όλα αυτά το κρατάει όρθιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν δείτε στις περισσότερο αναπτυγμένες περιοχές ε, μένει το 50% του ταμείου αυτού. Οπότε για να δούμε τις δυνατότητες του κοινωνικού ταμείου έχει σημασία με αυτό το οποίο είπατε να το συνδέσουμε, δηλαδή με τις υπηρεσίες, με θέματα αγοράς εργασίας, έτσι ώστε ο κόσμος να παραμείνει περισσότερο στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν σημαντικά μηνύματα λοιπόν ότι οι κοινωνικές διαστάσεις σε αυτή την περίοδο κρίσης δεν έχουν αρχίσει να σβήνουν αλλά λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε ότι σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε εξετάσει προσεκτικά το πλαίσιο στο οποίο αναφερθήκαμε και το κοινό στρατηγικό πλαίσιο το οποίο είναι σημαντικό για την ε, εφαρμογή. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού δεν θα πρέπει να υπάρξει μια απλή καταξουσιοδότηση πράξη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί τίθενται θέματα εδώ σημαντικά όπως η διαφάνεια, η λειτουργικότητα και δεν μπορούμε εμείς ε, ε, με μία θα έλεγα διατύπωση να τα ξεπεράσουμε. Απαιτείται μία συνομοθετική προσπάθεια. Έχουμε την αίσθηση, την πεποίθηση ότι θα ακολουθήσει τη συγκεκριμένη κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι θα μας καλύψει. Μετά το θέμα της εταιρικής σχέσης και είναι καλό σε επίπεδο κρατών μελών να μπορείτε να φτιάξετε θα έλεγα μία μια θέση στον τομέα σαν παράδειγμα της φροντίδας της υγείας η οποία ε, η θέση να ανταποκρίνεται στα επιμέρους χαρακτηριστικά και προβλήματα όλα αυτά θα πρέπει εμείς την πολιτική αυτή να τη διαμορφώσουμε εκ των κάτω προς τα πάνω για το 12 και το 13 σε συνεργασία με το κράτος μέλος, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, στα πλαίσια της περιφερειακής μας στρατηγικής. Για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε στη στρατηγική του 2020 και τους στόχους στην πολιτική συνοχής. Λοιπόν, δεν μιλάμε για πλήρη επανεθνικοποίηση, απλά μιλάμε για την συνεργασία του κράτους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρούμε λοιπόν και ελπίζουμε να υποστηριχθούμε από τα κοινοβούλια των κρατών μελών ότι θα μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να εφαρμόσουμε αυτήν τη νέα μέθοδο η οποία δεν θα οδηγήσει στην επανεθνικοποίηση. Τώρα η προσημείωση και ε, δεν νομίζω ότι στο τέλος θα πρέπει να καταλήξουμε με ένα δίσκαμπτο σύστημα χωρίς καμία ευελιξία. Νομίζω ότι σε σχέση με τα λειτουργικά προγράμματα θα μπορέσουμε να έχουμε τέτοιες λύσεις οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στα τοπικά χαρακτηριστικά και δεν θα εμείνουμε σε προκαθορισμένα ποσοστά και σε προκαθορισμένες θέσεις. Λοιπόν, χαίρομαι που είστε όλοι εδώ και συμμετέχετε σε αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω ότι με τη συζήτηση θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της οποίας όμως πρότασης η βάση είναι αποδεκτή. Dziękuję bardzo. I proszę o zabranie głosu. Ευχαριστώ. η κυρία Λούκα Σέβιτσα από το Λετωνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, πρόεδρε. Φυσικά πριν θέλω πρώτα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Πολωνικό Κοινοβούλιο για την διεξαγωγή αυτή τη συνάντησή μα, τη συνεδρίασή μα και για την επιλογή των θεμάτων. Οι πολίτε της Ευρώπης και η ευημερία της Ευρώπης είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μακροπρόθεσμα λοιπόν η ευημερία αηφόρος πολιτική για την απασχόληση είναι πάρα πολύ σημαντικές προϋποθέσεις σε περίοδο κρίσης. Η πολιτική για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης η 2020 απαιτεί προσπάθειες. Ακριβώς ε, από πλευράς της πολιτικής συνοχής πρέπει να διασφαλιστούν τα κονδύλια και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να διασφαλιστεί αυτή η συνάφεια, αυτή η διασύνδεση μεταξύ συνοχής και επαρκούς χρηματοδότησης. Κάνουμε λόγο για την κοινωνική συνοχή και για την ανάπτυξη των περιφερειών και περιοχών της Ευρώπης. Θέλουμε την παιδεία εκπαίδευση κατάρτιση να τονίσουμε και να τονίσουμε τη σπουδαιότητα των μέτρων στήριξης που έχουν μεγάλη σπουδαιότητα για την περιφερειακή ανάπτυξη θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω ότι πρέπει περισσότερα να επενδύσουμε στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και περιφέρειες. Από το 1995 ε, έως το 2005 στην Λετωνία και στη, χάρη στις προσπάθειες ε, ε, και τις επενδύσεις που έγιναν, οι περιφέρειες μας ε, κατάφεραν να ακολουθήσουν μια επιταχυμένη ανάπτυξη, μια ταχύ ανάπτυξη. Είμαστε σε θέση να ασφαλίσουμε αύξηση του ΑΕΠ από πλευράς Λετωνίας και διασφαλίστηκε το κοινωνικό κεφάλαιο όσον αφορά την παραγωγικότητα και το ΑΕΠ που αυξήθηκαν και η παραγωγικότητα και το ΑΕΠ όπως αυξήθηκε και η απασχόληση μέχρι την κρίση που μας έπληξε τώρα πρόσφατα και έτσι διαφοροποιούμαστε μεταξύ των πιο ισχυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πιο αδύναμων. Και αυτό δημιουργεί κινδύνους για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίοδο μετά την κρίση, της κρίσης και μετά την κρίση. Οι τάσεις που προανέφερα θα έχουν πολιτικές συνέπειες και επιπτώσεις. Η κοινωνική συνοχή από το 2,5% για παράδειγμα του ΑΕΠ ε, ως ε, ποσοστό. Δεν μπορούμε να δεχθούμε την πρόταση αυτή αυτής της διαφοροποίησης, διότι για τη Λετωνία θα σήμαινε αυτό 20% μείωση της, ε, των προπληρωμών και των προκαταβολών. Είναι μια μείωση πάρα πολύ αρνητική για την περίοδο της κρίσης και μετά την κρίση. Οι ίδιες οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζονται στην αλληλεγγύη και για την κοινωνική πολιτική και για την πολιτική συνοχή. Βασιζόμαστε στην αρχή της αλληλεγγύης. Πρέπει να έχουμε μια οικονομία που θα εδράζεται, θα βασίζεται σε αυτούς τους πυλώνες. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο και είναι οι πιο ευάλωτες να πληγούν ακόμα περισσότερο και να ακολουθήσουν ε, πολιτική αυστηρής λιτότητας και περικοπών. Πρέπει ε, να ακολουθήσουμε μια πολιτική σταθερής ανάπτυξης. Πρέπει να παραμείνουμε στα ίδια επίπεδα συγχρηματοδότησης που θα διασφαλίζονται. Δεν πρέπει να υπάρχουν αρνητικές διακριτικές, ε, αρνητική διακριτική μεταχείριση εις βάρος ε, των χωρών που είναι πιο αδύναμες, ιδιαίτερα όσον αφορά την πολιτική αλληλεγγύης και συνοχής θα πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό εκφράζω την ελπίδα ότι κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων και μετά από αυτές για την ανάπτυξη και εξέλιξη της πολιτικής συνοχής θα βασιζόμαστε και θα εκφραζόμαστε με τις αρχές που εκφράζουμε την αρχή της αλληλεγγύης που πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή με αυτόν τον τρόπο που θα διασφαλίζεται. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και χώρες να υποστηριχθούν περισσότερο. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία θα διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό χαίρομαι για το ότι μπορούμε να συζητήσουμε με αυτόν τον τρόπο και να ανταλλάξουμε απόψεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να εκφραστώ ενώπιον σας. Ελπίζω σε επικοδομητικές συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Από την Πολωνική Γερουσία ο κύριος Βίτμπολτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που ανέφερε η κυρία Κρέλη, η συγγήτρια σχετικά με τις δημογραφικές προκλήσεις και προσδιορίζοντας δύο μέσα, τη στρατηγική 2020 και την πολιτική συνοχής. Πρόκειται για μέσα κλειδί, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό, κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, αφορά το επίπεδο της Ένωσης και τη στρατηγική για την ευφύ ανάπτυξη και την κοινωνική συμπερίληψη που υλοποιείται στα διάφορα κράτη-μέλη και μετά έχουμε το επίπεδο των κρατών μελών για το οποίο μιλήσαμε πολύ στο πάνελ. Μιλήσαμε για την εργασία, για τη συνταξιοδότηση, ηλικία συνταξιοδότησης, για την υγιεινή στο χώρο εργασίας. Αυτά όλα είναι όμως σε εθνικό επίπεδο. Εκείνο που θεωρώ εγώ το πιο σημαντικό είναι το περιφερειακό επίπεδο, γιατί ό,τι έχει να κάνει με τη συνοχή πρέπει να υλοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο. Όπως είπε ο Λιθωνός συνάδελφος, είναι τεράστια η δυναμική των περιφερειών. Η συνοχή εξαρτάται όμως από διάφορους παράγοντες από την οικονομία της, από την περιφέρεια, από τη δημογραφική της ανάπτυξη και διαφέρουν όλοι αυτοί οι παράγοντες. Γι' αυτό η χρηματοδότηση υπέρ της πολιτικής συνοχής εξαρτάται ως προς την επιτυχία της από το πώς λειτουργούν και πράττουν οι περιφέρειες. Για μας τους Πολωνούς η πολιτική συνοχής πρέπει, είναι αποτελεσματική αλλά πρέπει να δοθεί διαφορετική απάντηση ανάλογα με την περιφέρεια στην Ευρώπη. Πρέπει να κάνουμε και μια πολιτική αναβάθμιση αυτής της πολιτικής. Τα κονδύλια της συνοχής θα πρέπει να διατηρηθούν στα ενά επίπεδα, αν, ε, αν όχι να αυξηθούν. Έχουμε το Eurofencing, έχουμε την European Connecting Facility, ε, που εντάσσονται σε όλα αυτά τα επίπεδα. Όλα αυτά δεν θα πρέπει να υπονομεύσουν τα δεδομένα στα οποία έχουμε καταλήξει σήμερα και τις κατακτήσεις τις οποίες έχουμε καταλήξει σήμερα. Σας ευχαριστώ κύριε Γερουσιαστά. Όποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο παρακαλώ να συμπληρώσει το μικρό έντυπο και να το καταθέσει. Ο κύριος Νούνιο έχει το λόγο από την Πορτογαλική Βουλή. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Μπορεί να υπάρχει κοινωνική συνοχή και εφόρος ανάπτυξη με ισορροπία για την ίση και δίκαιη ανάπτυξη των περιφερειών. Στην Πορτογαλία εδώ και χρόνια παρουσιάζεται μια τάση μετανάστευσης ε, του πληθυσμού από το εσωτερικό στις παράκτιες περιοχές αναζητώντας ε, και την απασχόληση σε μεγάλες πόλεις. Αυτό το φαινόμενο οδηγεί στην αποψήλωση του εσωτερικού, της εσωτερικής χώρας, ε, της της Μεσογείου χώρας, προς τα οικονομικά κέντρα. Δημιουργούνται προβλήματα ανεργίας στις ε, μεγάλες πόλεις ε, και αποψηλώνονται οι περιοχές όπου μόνο μένουν οι γέροι που ζουν σε αυτές. Ε, έχουμε ανισορροπίες δημογραφικές και έχουμε μια, ένα πληθυσμό νεότερο από πλευρά ηλικία τη πόλη. Έχουμε και τη διαφορετική μορφή ζωής που ε, δεν δίνει δυνατότητα να ευδοκιμήσουν όλες, όλοι οι στόχοι. Έχουμε λοιπόν την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι σωστές ισορροπίες. Ένα άλλο πρόβλημα είναι στην περίοδο κρίσης και πολιτικών λιτότητας δημιουργείται η ανάγκη να επιλέγονται πολιτικές πιο κεντροσχεδιασμένες, ε, ε, κεντρική σχεδίασης. Στην Πορτογαλία δυστυχώς ε, υπάρχει ακόμα ιδέα ότι η αποκέντρωση και η μεταφορά αρμοδιοτήτων και κονδυλίων για τις περιφέρειες μπορεί να σημαίνει μια μεγαλύτερη, ας το πω έτσι, διαμόρφωση κινδύνων όσον αφορά την περίοδο κρίσης. Αυτό τον κίνδυνο πρέπει να τον απομακρύνουμε. Πρέπει να μην πέσουμε σε μια παγίδα αυτού του είδους. Έτσι η περιφερική ανάπτυξη είναι ένα στίχημα που πρέπει να κερδίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες προκλήσεις, αλλά να διατηρείται πάντα στους κεντρικούς άξονες ε, που προσανατολίζουν τις πολιτικές μας. Πρέπει να έχουμε τα επίπεδα ανάπτυξης ε, για την επίτευξη εξυγχρονισμού μιας ε, μεγάλης ένωσης όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να ενδυναμωθεί και μπορεί να δώσει κίνητρα να αυξηθούν τα ποσοστά γεννητικότητας με τις νέες ευκαιρίες που θα δημιουργούνται για ολόκληρο τον πληθυσμό. Ευχαριστώ. Ε, e, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Χίμπνερ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιας και δεν υπάρχουν περισσότεροι που έχουν ζητήσει το λόγο και πριν δώσω το λόγο στην κυρία Κρέλ θα ήθελα να σας ενημερώσω σαν πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για κάποια από τα θέματα τα οποία συνδέονται με τις εργασίες μας και με το μελλοντικό διακανονιστικό πλαίσιο. Τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε πιο ισχυροί στα πλαίσια της συναπόφασης με το Συμβούλιο για τη μελλοντική μορφή την οποία θα πρέπει να πάρει η συνοχή, η πολιτική συνοχής και η πολιτική περιφερειακή. Αυτό σημαίνει ότι νιώθουμε και περισσότερο υπεύθυνοι από ό,τι στο παρελθόν. Τα τελευταία δύο χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πάρει συγκεκριμένες θέσεις για τη χρηματοδότηση των μελλοντικών πρόπτικων. Έχει πάρει αποφάσεις μέσω εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας της Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσπαθώντας να κατανοήσουμε το περιεχόμενο των μελλοντικών προτάσεων και συμμεριζόμενοι με το Συμβούλιο και την Επιτροπή τις ίδιες αξίες και τους ίδιους πολιτικούς στόχους. Μπορώ λοιπόν να πω ότι η συγητής μας και η Περιφερειακή μας Επιτροπή είναι πλέον προπαρασκευασμένοι να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατόν. Πρόθεσή μας, όπως γνωρίζετε, και είναι και η πρόταση της ε, Τρόικας της Προεδρίας, να προσπαθήσουμε να συμπληρώσουμε την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει για το επόμενο διακανονιστικό πλαίσιο μέχρι το τέλος του 12. Θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω ότι κάτι τέτοιο θα εξαρτηθεί επίσης και από το πώς οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα προχωρήσουν. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, διαπραγματευόμενοι το διακανονιστικό πλαίσιο μπορούμε να προτείνουμε κάποιους αριθμούς οι οποίοι να είναι σε εισαγωγικά, αλλά χωρίς αριθμούς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Πάρα πολλά και πάρα πολλές λύσεις για το μέλλον θα εξαρτηθούν από τις διαθέσιμες πιστώσεις. Θα πρέπει να πιέσετε λοιπόν και εσείς τις κυβερνήσεις σας έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα πλαίσια του νέου διακανονιστικού πλαισίου στον επόμενο προϋπολογισμό για να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Το Κοινοβούλιο δεν θα επιβραδύνει τη διαδικασία και να μην ξεχάσετε ότι υπάρχει και ο δικός σας ρόλος, τον οποίο θα εκτιμήσουμε ιδιαίτερα, και οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλοι έχουμε την πολιτική ευθύνη είτε σαν συμπολίτευση είτε σαν αντιπολίτευση και στο Κοινοβούλιο και στις ε, χώρες μέλη να επηρεάσουμε τις απόψεις των κυβερνήσεών μας. Ο ρόλος σας θα πρέπει να πηγαίνει και πέραν των περιοριστικών μέτρων και των μέτρων ε, δημοσιονομικής πειθαρχίας που λαμβάνονται μέχρι τώρα θα πρέπει και εσείς πιο μακροπρόθεσμα να κατανοήσετε ότι απαιτείται ανάπτυξη στην Ευρώπη και για να το πετύχουμε αυτό απαιτείται ένας επαρκής προϋπολογισμός ο οποίος θα μας επιτρέψει να επενδύσουμε στους τομείς όπου κάτι τέτοιο χρειάζεται. Και αναφέρομαι εδώ στον ρόλο των πόλεων, στον ρόλο των περιφερειών, των περιοχών, Να σας ενημερώσω επίσης ότι τα τελευταία χρόνια οργανώσαμε και πάρα πολλές ακροάσεις. Συζητήσαμε με πάρα πολλούς εμπλεκόμενους έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις τις οποίες παρουσιάζει το παρόν σύστημα και πώς οι εισηγητές μπορούν να λάβουν καλύτερα υπόψη τους αυτά τα οποία ακούγονται από τη βάση. Να σας πω επίσης ότι μιας και βρίσκεστε εδώ, να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία τροποποίησης του ισχύοντος κανονισμού λόγω της κρίσης μετά από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα χρήματα. Μία από τις τροπολογίες, η οποία ήδη ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, αφορά την αύξηση, το λεγόμενο top-up. Μια άλλη τροπολογία αφορά τα θέματα του λεγόμενα του financial engineering, Νομίζω ότι και εκεί θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάποια λύση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα πλαίσια του μέσου ε, διασποράς του κινδύνου, έτσι ώστε και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να σταθεί πιο χρήσιμη από ό,τι σήμερα. Ιδιαίτερα σε μία περίοδο υψηλού δημοσίου χρέους. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εμείς υπολογίζουμε στη δική σας συνεργασία, στη δική σας προσπάθεια. Είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην προσπάθεια αυτή και τώρα και για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον Μίετσεσλάβ Αουγκούστιν της Πολωνικής Γερουσίας. εξετάζουμε την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά μέσα από μια ιδιάζουσα οπτική, δηλαδή τις επιπτώσεις που όπως προκύπτουν από τις δημογραφικές αλλαγές που διαμείβονται στην Ευρώπη σήμερα. Στο προηγούμενο πάνελ είπαμε ότι η κατάσταση διαφέρει ιδιαίτερα από κράτος σε κράτος ή από περιφέρεια σε περιφέρεια κάθε κράτους μέλους. Φυσικά, το να εξαλείψουμε τις διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών θα βελτιώσει και την κοινωνική κατάσταση αυτών των περιφερειών και πιο συγκεκριμένα την κατάσταση των ηλικιωμένων. Υπάρχουν όμως τομείς στην πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης που δημογραφικά από δημογραφικής πλευράς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις πιο επικίνδυνες περιοχές, ε, τις περιοχές που, που ρηψοκινδυνεύουν την γύρανση, από τη γύρανση του πληθυσμού. Μιλάω εδώ για επενδύσεις, απαραίτητες επενδύσεις σε υγειονομικές υποδομές και κυρίως ε, στην πρόληψη. Αν θέλουμε οι ηλικιωμένοι να εργάζονται περισσότερα χρόνια πρέπει να είναι και πιο υγιείς. Στο προηγούμενο πάνελ υπόθηκε ότι σε ορισμένες χώρες όπως η Εστονία και η Ουγγαρία η κατάσταση είναι κατεπίγουσα. Διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τέτοιες υγειονομικές συνθήκες δεν μπορούν να, για να εργάζονται για πολύ καιρό. Και αφήστε δε και την αποκατάσταση. Δηλαδή αν ένας ε, ηλικιωμένος μετά από ένα δυστύχημα πρέπει να ξαναρχίσει να, να, να, δουλεύει, ε, θα πρέπει να αποκατασταθεί. Δηλαδή έχουμε κάθε συμφέρον να αποκατασταθεί για να συνεχίσει να δουλεύει και να μην βγει στη σύνταξη. Και υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις υποδομών για την αποκατάσταση. Υπάρχουν δύο ταχύτητες ε, στην γύρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Αφενός έχουμε την κατηγορία πάνω από το 80, μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα για, τα, για οποία ε, με το, για το, δεν μπορεί να ασχοληθεί η οικογένειά τους. Και στην Ευρώπη είμαστε καταδικασμένοι όλοι να τύχουμε αυτή της βοήθειας. Πού βρίσκεται όμως αυτή η βοήθεια, σε ποιες περιοχές, πώς θα πρέπει να επενδύσουμε σε επίπεδο περιφερειακής πολιτικής. Και έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε και νέες θέσεις εργασίας. Ένα άλλο ζήτημα είναι το θέμα της εκπαίδευσης, όχι μόνο για τους νέους, αλλά και για τους ηλικιωμένους. Η δουλειά είναι συνεχώς πιο απαιτητική και συνεχώς πιο μηχανική, πιο, πιο μηχανογραφημένη. Χρειάζεται λοιπόν κατάρτιση για τους ηλικιωμένους μια δεύτερη, τρίτη ευκαιρία. Και εδώ πάλι οι διαφορές είναι μεγάλες ανάλογα με το κράτος μέλος και τις περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν όταν εμείς ψάχνουμε τα, σχέδια, τα διάφορα σχέδια, αναλύουμε τα σχέδια και τους διάφορους στόχους, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία, διότι εδώ είναι η προπτική της ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών. Ευχαριστώ κύριε Γερουσιαστά. Κύριες και κύριοι, τώρα δίνω την Προεδρία στην κυρία Ντανούτα Χιούμπνερ. Έχετε το λόγο. Ως ε, πρόεδρος ε, θα δώσω και πάλι το λόγο στην κυρία Κρέλ. Θα περιοριστώ δηλαδή σε αυτό για να σχολιάσει η κυρία Κρέλ ε, τα διάφορα, τις, τις διάφορες τοποθετήσεις των συναδέλφων του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Κρέλ. Äh, Ευχαριστώ κύριε, κυρία Πρόεδρε. Διαπιστώνω ότι στα εθνικά κοινοβούλια συζητάτε ακριβώς τα ίδια πράγματα που συζητάμε εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παντού οι απορίες είναι οι ίδιες, πώς θα αναπτυχτούμε, προς τα πού θα τίνουμε. Σε όλα τα επίπεδα λοιπόν είναι αντίστοιχες οι σκέψεις και οι προβληματισμοί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συστήσει μία ειδική υποεπιτροπή για τις δημοσιονομικές πρόπτικες από το 2014 και μετά. Πρόκειται για την περίφημη έκθεση Γκαρίγκα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι είπε ότι αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί αν θέλουμε να απαντήσουμε στις προσδοκίες των περιφερειών, ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 5%. Και αυτό υπόθηκε σε μια, σε μια φάση κρίσης, κρίσης που εξάλλου υφίσταται ακόμα. Αυτό το οποίο πρότεινε βέβαια η Κομισιόν είναι χαμηλότερο από αυτό που πρότεινε το Κοινοβούλιο και ακόμη και με το Connecting for Europe έχουμε μόνο 326 εκατομμύρια για τα ταμεία συνοχής, δηλαδή βγάζοντας το Connecting Europe. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μία λύση. Η Κομισιόν πρότεινε λίγα πράγματα και αυτά τα οποία πρότεινε η Κομισιόν δεν έγιναν ακόμη δεκτά από το Συμβούλιο. Ακόμη δηλαδή και γι' αυτό το μικρότερο ποσό θα γίνουν μεγάλες συζητήσεις, ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται από τις ε, διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό και στις χώρες σας. Δηλαδή σας δίνουν κάτι από τη μια μεριά, αλλά για να το πάρετε πρέπει να διαγράψετε μια δαπάνη κάπου αλλού. Πού θα τα βρούμε όμως αυτά τα χρήματα, πού θα τα κόψουμε. Εγώ σας παρακαλώ σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να υποδείξετε προς τους υπουργούς οικονομίας ότι αξίζει τον κόπο να επενδύσουν σε μια πολιτική συνοχής. Διότι η συνοχή είναι προς το κοινό συμφέρον όλων και για τους λιγότερο ανεπτυγμένους και για τους περισσότερο αναπτυγμένους. Θα πρέπει να επιμείνετε στις περιφέρειές σας και στις χώρες σας, ούτως ώστε να ασκηθούν πιέσεις, ώστε να καταλήξουμε σε μία ισορροπία μεταξύ των περιφερειών που είναι δικαιούχοι του χρήματος και των χωρών που χρηματοδοτούν. Αυτή την ισορροπία ακόμη δεν την έχουμε βρει και διατρέχουμε τον κίνδυνο να δημιουργήσει ακόμη προβλήματα και δύσκολες διαπραγματεύσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα στρατευμένο προς αυτήν την κατεύθυνση και... Θέλουμε να το παλέψουμε στη συνέχεια των συζητήσεών μας, διότι βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Στην τελευταία Ολομέλεια εγκρίναμε μία έκθεση για τη δημογραφική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επιπτώσεις της πολιτικής συνοχής και διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Και άμα δείτε και τις διάφορες προτεραιότητες που προτάθηκαν και κυρίως αυτές ε, οι οποίες ε, ε, σχετίζονται με τις πολιτικές σύνοχης και αν σας πω ότι θέλουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα σε τεχνολογικό επίπεδο για την επικοινωνία, την πληροφόρηση. Αυτό πρέπει να γίνει παντού, πρέπει να γίνει σε όλες τις περιφέρειες. Θα πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση και να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις νέες τεχνολογίες εχμής. Και φυσικά και πιο ηλικιωμένοι θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνία της πληροφόρησης. Τώρα όταν λέμε επίσης ότι θέλουμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα πρέπει όμως να βοηθήσουμε όχι μόνο τις μεγάλες χαλιβουργίες, θα πρέπει να βοηθήσουμε και τις ε, μικρομεσαίες εκείνες επιχειρήσεις οι οποίες εργάζονται στον τομέα της υγείας. Και όταν λέμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτελεσματικότητα της ε, χρήσης των φυσικών πόρων. Αυτό ισχύει για όλες τις περιφέρειες. Περιφέρειες είτε με μεγάλο είτε με μικρότερο πληθυσμό, υποδομές επίσης στις μεταφορές. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έχουμε έναν πληθυσμό που θα γερνάει όλο ένα και περισσότερο. Θα πρέπει να ξέρουμε κυρίως όσον αφορά στις αστικές περιοχές ποιοι θα είναι οι χρήστες των μαζικών μέσων συγκοινωνίας για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε αυτά τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας στις ανάγκες του πληθυσμού. Και αν έχω εγώ έναν πληθυσμό ο οποίος όλο ένα μειώνεται στην περιφέρεια, μήπως δεν θα έπρεπε να αλλάξω το σύστημα των υποδομών μου. Έχετε επίσης την διαβίου κατάρτιση και αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποτελεί μία από τις προτεραιότητές μας. Αλλά αν λάβουμε υπόψη αυτές τις 11 προτεραιότητες που βρίσκονται στο βασικό κανονισμό, θα πρέπει αυτές τις προτεραιότητες, να τις δούμε με μια σχετική ευελιξία που θα λαμβάνει υπόψη την μείωση του πληθυσμού. Το δημογραφικό πρόβλημα, να δούμε αν θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε ορισμένα σημεία βασισμένοι σε συμβόλαια κατάρτισης προτεραιοτήτων. Για τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές θα μπορούσαμε να είχαμε έναν κατάλογο επιλογών, για τις άλλες όμως όχι απαραίτητα οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ξέρω ότι στην Ισπανία έχετε ορισμένες περιοχές οι οποίες είναι εντελώς ε, απεριμωμένες σήμερα και χρειάζεται να τις ε, προσεγγίσουμε με μια διαφορετική οπτική από ότι οι παραλιακές περιοχές. Εγώ έρχομαι από την Ανατολική Γερμανία και στην Ανατολική Γερμανία έχουμε περιοχές οι οποίες έχουν μείνει χωρίς νεολαία, διότι δεν υπήρχε δουλειά. Οπότε φύγανε. Πρέπει να προβλέψουμε κατά συνέπεια πώς θα θέσουμε στην υπηρεσία των ηλικιωμένων νέες υποδομές. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα γύρω από την αρχή της αιρεσιμότητας. Πρέπει να βρούμε ένα σύστημα το οποίο να λειτουργεί πραγματικά. σε επίπεδο προτεραιοτήτων πάντα στα πλαίσια των συμφωνιών συνεργασίας θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις υποδομές στα πλαίσια των υποδομών. Είναι ένα θέμα το οποίο θέλουμε να διαπραγματευτούμε με την Κομισιόν. Σχεδόν όλοι υπογράμμισαν και το πόσο σημαντική είναι η επαγγελματική κατάρτιση και για τους νέους και για τους λιγότερο νέους. Όπως επίσης και την διάθεση όλων των υποδομών που συνδέονται με αυτή την κατάρτιση. Πρόκειται για ένα άλλο ζήτημα γύρω από το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί το Κοινοβούλιο και να δούμε πώς θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια τα οποία θα είναι αναγκαία να δοθούν στις αναγκαίες υποδομές που πρέπει να δημιουργηθούν. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό, θα έλεγα, για την επόμενη περίοδο σχεδιασμού από το 2014 μέχρι το 2020 και από το 2014 στο 2020 επαναλαμβάνω. Και θα παρακαλούσα λοιπόν και ίσως θα μπορούσαμε με σχόλια και απόψεις που θα μας διαβιβάσετε να δούμε και να ξανασκεφτούμε αν το αποθεματικό αυτό επιδόσεων θα μπορούσε να βοηθήσει. Δεν είναι ότι το 5% κάπου στις Βρυξέλλες θα βρίσκεται και θα έρχεται κάποιος και θα λέει πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια, όλοι οι στόχοι μπορούν να, μια και έχουν επιτευχθεί να γίνουν, να πάνε και πιο πέρα. Αν μέλος είναι το 5% αποθεματικού επιδόσεων που διατηρείται. Δεν θα είναι μια νέα ανακατανομή κονδυλίων, αλλά πραγματικά στα ίδια τα κράτη-μέλη θα μπορεί αυτό να είναι κίνητρο, ώστε περισσότερη δημιουργικότητα και με πιο ευφυή τρόπο οι περιφέρειες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κίνητρα. Αν έχουν δουλέψει και έχουν, κάνει, έχουν καλές επιδόσεις θα μπορούν να επιστρέψουν και να πάρουν επιπρόσθετα κονδύλια για να συνεχίσουν το θετικό έργο. Θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι από κοινού. Θα ήταν ένα ευφυές έργο μετά από όλους τους όρους και προϋποθέσεις ερεσιμότητας όταν λένε όλοι το ένα δεν επιτρέπεται, το άλλο δεν επιτρέπεται. Πρέπει να έχεις όρους και προϋποθέσεις να έχουμε κίνητρα ώστε με τα κίνητρα να μπορέσουν να προχωρήσουν τα πιο θετικά προγράμματα και ε, ε, σχέδια με τις βέλτιστες ε, προδιαγραφές με τις βέλτιστες ε, επιδόσεις να μπορούν να προχωρήσουν. Πώς θα μπορούσε το μέσο για τη διασύνδεση και ε, ένωση της Ευρώπης, Connecting Europe, να προχωρήσει. Έχουμε έντονες συζητήσεις που διεξάγονται και στις χώρες μας. τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα έχουμε σε βάθος επαφές μαζί σας, θα εμβαθύνουμε τις επαφές μαζί σας και με τα κράτη-μέλη, ώστε να προχωρήσουμε πιο πέρα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτή την εξέλιξη, προς αυτή την πορεία. Ελπίζω όλα τα θέματα τα οποία αναφέρατε καλύφθηκαν και χαίρομαι πραγματικά για μια καλή συνεργασία, θετική, επικοδομητική συνεργασία. Αν έχετε κάποιες προτάσεις που θέλετε οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη σε αυτόν τον κανονισμό, σε αυτό το νομοθετικό πακέτο μέτρων, είμαστε συνομοθέτες, είμαστε ακριβώς σε αυτή τη φάση διατύπωσης των κανονισμών, των προδιαγραφών του κανονισμού τότε στείλτε μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις απόψεις σας, ώστε από κοινού να σημειωθεί πρόοδος στις διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική πολιτική συνοχή και να ξανασυζητηθούν όλα αυτά. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, thank you very much. Σας ευχαριστώ, Κωνσταντσε Κρέλ θα ήθελα να ζητήσω από τον δεύτερο σχολιαστή, εισηγητή μάλλον, τον κύριο Φανίστεν Ρόι να συμπληρώσει κάτι. Θα είμαι σύντομος, λέει ο κύριος Βανρίστερ Ρόι. Ένα πράγμα, ίσως ε, περιθωριακό να ακούγεται για κάποιους. Την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πολιτική της στον τομέα της έρευνας Η έρευνα αυξάνεται από 54 δις σε 80. Αλλά βλέπουμε ότι το 90% από τα χρήματα αυτά πηγαίνει στα λεγόμενα παλαιά κράτη-μέλη. Άνω του 90% δίδεται σε πανεπιστήμια και σε επιχειρήσεις στις παλιές λεγόμενες χώρες. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν εμείς να προσαρμόσουμε τις δυνατότητές μας και στα νέα κρατημέλη για να μπορέσουν τα νέα κρατημέλη να γίνουν ανταγωνιστικά και για την έρευνα. Τα χρήματα αυτά δίδονται σε αυτούς οι οποίοι πράγματι ε, μπορούν να τύχουν αριστείων για την προσπάθεια την οποία κάνουν και γι' αυτό θα πρέπει στην περίοδο 2014 με 2020 να βελτιώσουμε την πρόσβαση αυτή προς την αριστεία και μέσω των πολιτικών συνοχής. Μπορεί κανείς να δαπανίσει περισσότερα χρήματα δημιουργώντας υποδομές για την έρευνα, εκεί όπου χρειάζεται βέβαια, εκεί που υπάρχουν δυνατότητες ακαδημαϊκές πανεπιστημιακές, να είναι κανείς ικανός και να βοηθείτε για να γίνει περισσότερο ικανός. Αυτό είναι πράγματι ο δρόμος για την αριστεία. Όταν ήμουνα στην Πολωνία είχα συναντηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών και με τον Υπουργό τον Υπεύθυνο για την Εκπαίδευση και την Τεχνολογία και ακριβώς αυτό είχαν στο νου τους. Θα πρέπει λοιπόν η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πιο ισόρροπη γεωγραφικά μετά από μια κάποια τουλάχιστον περίοδο. Δεν ξέρω πώς θα χτίσουμε λοιπόν αυτό τον δρόμο προς την αριστεία, αλλά οφείλουμε να τον χτίσουμε. Ευχαριστώ Λάμπερ Βανίστεροι. Φτάνουμε στο τέλος της συζήτησης. Θα ήθελα εδώ για μια ακόμη φορά να πω δύο πράγματα. Πρώτον, τα επόμενα χρόνια θα βιώσουμε καταστάσεις περίεργες. Σας ελπίσουμε ότι θα είναι καταστάσεις μετά την κρίση. Η Ευρώπη λοιπόν θα χρειάζεται ανάπτυξη, απελπισμένα θα χρειάζεται νέους ρυθμούς ανάπτυξης. Ανάπτυξη η οποία αναβασίζεται σε διάφορους τρόπους, σε διάφορες μεθόδους, σε διάφορες πλατφόρμες, και ιδιαίτερα στον τομέα των κερδών στην παραγωγικότητα. Εάν πράγματι στην Ευρώπη θέλουμε να έχουμε σταθερές θέσεις εργασίας, θέσεις οι οποίες δεν θα χαθούν αύριο και θα πάνε σε άλλες αναδυόμενες οικονομίες, αυτές οι θέσεις θα πρέπει να βασίζονται σε μία ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι μπορούμε να δούμε ποιοι είναι οι τομείς που θα δώσουν ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Αυτό μπορεί να ποικίλει ανά περιοχή, μπορούμε να βρούμε διαφορετικά μέτρα στη Βουλγαρία ή στη Φιλανδία. Πρέπει όμως να έχουμε μια πολιτική η οποία να, μας να λαμβάνει υπόψη όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά των επιμέρους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο φτωχότεροι είμαστε στην ανταγωνιστικότητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια την οποία θα πρέπει να κάνουμε. Και θα πρέπει η καινοτομία να υποβοηθείται και όχι μόνο στις πλούσιες χώρες, αλλά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο. Εσείς γνωρίζετε τις περιφέρειές σας, γνωρίζετε τις πόλεις σας, τις επαρχίες σας, και πρέπει να ενθαρρύνετε αυτούς που έχουν δυνατότητες στις περιοχές σας και αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με την περιφερειακή πολιτική να προωθήσουν τις πολιτικές οι οποίες ε, είναι χρήσιμες. Εμείς ε, θα συναντηθούμε τον Οκτώβριο ε, του επομένου έτους ξανά, αλλά νομίζω ότι ήδη από πριν πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνούμε. Στους εισηγητές υπάρχουν όλες οι πολιτικές αποχρώσεις και οι πολιτικές ομάδες. Πάντα μπορείτε να εντοπίσετε ένα εισηγητή, ένα σκιώδη εισηγητή και εισηγήτρια και να μπορέσετε να συνεργαστείτε μαζί του. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και για να συνεργαστούμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για τη συνάντηση αυτή και ελπίζουμε η συνάντηση αυτή να γίνει μονιμότερη και να μην είναι μόνο μία εφάπαξ κατέτος συνάντηση. Να σας πληροφορήσω ότι θα υπάρξει μία μικρή δεξίωση πριν από το δείπνο. Προσπαθούμε να βάλουμε το δείπνο λίγο νωρίτερα, δεν έχω τα αποτελέσματα, αλλά παρακαλώ τώρα να κατεβείτε από, την κεντρική, από το κεντρικό κλιμακοστάσιο στην αίθουσα Γεχούντι Μενούχιν όπου θα σας περιμένουν ποτά και αργότερα θα ξεκινήσει εκεί το δείπνο. Ευχαριστώ.